να σας καλωσορίσω σε αυτή τη συνεδρίαση των Επιτροπών της Eurolat και να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Τα μέλη της ε, Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Eurolat, ε, τα μέλη του Διπλωματικού Σώματος, πρέσβεις που συμμετέχουν στην συνεδρίαση, ε, τους ειδικούς προσκεκλημένους, να τους ευχαριστήσω όλους και να γενιάσουμε τη συνεδρίαση αυτή ενημερώνοντάς σας ότι έχουμε διερμηνία σε πορτογαλικά, ισπανικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ε, και πολωνικά και ελληνικά οπότε θα περάσουμε κατευθείαν στην εναρκτήρια σύνοδο κατόπιν θα έχουμε ένα σύντομο διάλειμμα και στο τέλος θα ακούσουμε τη δήλωση της Μαρία Μεχία θα ακολουθήσει συζήτηση και στην ίδια αίθουσα θα κάνουμε και την οικογενειακή φωτογραφία ενώ το απόγευμα και πριν τη συνέντευξη τύπου θα συνεδριάσουν οι Έχουμε μαζί μας τον Επίτροπο Αντώνιο Ταγιάννη, τον Αχιλίνο Γκαρσόν, αντιπρόεδρο της Κολομβίας, την Μπενίτα Βάρκερ, πρόεδρο της του Ιδρύματος EULAC, την Αλίσια Μπάρσενα, εκτελεστική γραμματέα της ΕΚΛΑΚ e και την Γκλώρια Ορκελή, την πρόεδρο τη Λατινοαμερικανικής Συνιστώσης. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ταγιάννη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ των Λατιναμερικανικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που έχω την ευκαιρία να μιλήσω και εδώ μετά την ε, παρουσία μου στη Σεβίλη το 2010. Θα ήθελα ευθύ εξ αρχής να διακηρύξω ότι αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε και περισσότερη Ευρώπη και περισσότερη Λατινική Αμερική και στενότερη συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής. Σε αυτή τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής ο ρόλος των κοινοβουλίων είναι ουσιώδης. Θα πρέπει να συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε την οικονομική ανάπτυξη των υπήρων μας γιατί έχουμε κοινή ιστορία, θρησκεία, γλώσσες, πολιτισμό και ε, έχουμε πάθος για το ποδόσφαιρο και για παρόμοια αθλήματα. Και μάλιστα όταν άλλοι παγκόσμιοι ε, φορείς κατακλείζουν την παγκόσμια σκηνή, ε, θεωρώ ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος. Γιατί στην ε, Λατινική Αμερική έχετε 600 εκατομμύρια κατοίκους, 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Έχετε τεράστιο ρηκτό πλούτο και ενεργειακούς πόρους. Ταυτόχρονα και το πιο σημαντικό, έχετε ένα σημαντικότατο ανθρώπινο κεφάλαιο. Εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε 500 εκατομμύρια ψυχέ. Εδώ και 60 περίπου χρόνια ενισχύουμε και βαθύνουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Έχουμε μια ενιαία αγορά και εξακολουθούμε να είμαστε η πρώτη παγκοσμίω εμπορική δύναμη. Σε αυτή τη στιγμή όμω τη σοβαρή χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση στην Ευρώπη, μερικέ τρίτε χώρε μα αντιμετωπίζουν κάπω υπεροπτικά. Θεωρούν ότι είμαστε εξοφλημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη. Εγώ διαφωνώ με τη γνώμη αυτή. Σίγουρα η Ευρώπη θα βγει πολύ διαφορετική από την κρίση που διανύει. Αλλά πιστεύω ότι η Ευρώπη θα βγει από την κρίση αυτή πιο ισχυρή, πιο συνεκτική και ακόμη πιο ανταγωνιστική. Νομίζω ότι είναι προς συμφέρον και των δύο υπήρων να είναι ισχυρότερη η Ευρώπη, πιο συνεκτική και πιο ανταγωνιστική. Δεν πρόκειται να σας κατακλείσω με αριθμητικά στοιχεία. Θα σας δώσω μόνο λίγα νούμερα. Οι Ευρωπαϊκή επενδύσεις στη Λατινική Αμερική είναι τριπλάσιες από τι αντίστοιχε ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Κίνα, την Ινδία και τη Ρωσία μαζί. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να μας θάψουν πριν την ώρα μας. Εργαζόμαστε σκληρά για να δώσουμε νέα πνοή στις διαπραγματεύσεις του Μερκοσούρ και σε άλλες παρόμοιες διαπραγματεύσεις. Σας διαβεβαιώ ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις δικές μου αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει ζωηρό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για τη Λατινική Αμερική. Είναι πολύ σημαντική συνεργασία με τη Λατινική Αμερική σε θέματα εξωτερικής πολιτικής ε, και εμπορικής πολιτικής. Πάντως προσπαθώ να δώσω έμφαση και σε ένα τρίτο πεδίο συνεργασίας μεταξύ μας. Να συμπληρώσουμε την εξωτερική πολιτική και την εμπορική πολιτική με επιχειρηματική και βιομηχανική συνεργασία. Γι' αυτό και μετέβη στη Χιλή, την Αργεντινή και τη Βραζιλία τον περασμένο Ιούνιο. Ε, πάνω από 15 χρόνια είχα περάσει πριν ένας ε, επίτροπος βιομηχανίας και επιχειρήσεων πραγματοποιήσει επίσκεψη στην περιοχή και μάλιστα σε τρεις εβδομάδες ε, θα πάω στη Βραζιλία και στην Αργεντινή όταν μου επιτρέψει το πρόγραμμά μου. Αυτή τη στιγμή θα πάω μόνο στη Βραζιλία. Δεν θα πάω μόνος μου στη Βραζιλία. Θα με συνοδεύσει ένα σημαντικό επιτελείο εκπροσώπων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Είναι σημαντικό ότι ε, και οι τοπικοί ηγέτες συνοδεύονται με επιχειρηματίες στα ταξίδια τους στην Αλοδαπή. Το σχέδιο μου αυτό είναι καινοτόμο γιατί δεν ήθιστε ένας πολιτικός από την Ευρώπη να συνοδεύεται από Ευρωπαίους επιχειρηματίες. Θα με συνοδεύσουν περίπου 20 ε, άνδρες και γυναίκες που είναι διευθυντές σημαντικών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Θέλουμε να δείξουμε από κοινού το ενδιαφέρον μας για τη Βραζιλία και όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το Μερκοσούρ, νομίζω ότι μπορούμε να συμβιώσουμε πρόοδο σε σημεία κοινού ενδιαφέροντος. Ε, βέβαια, από τα σημαντικότερα θέματα είναι η πρόθεση των ε, ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το 13% έχουν εξαγωγέ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάτι που είναι ανεπαρκές, ένα πολύ αμεληταίο ποσοστό. Και μάλιστα τη στιγμή που έχουμε πολύ χαμηλή οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνουμε μία έξοδο. Πρέπει να ενισχύσουμε τις εξαγωγές μας προς τη Λατινική Αμερική. Κατά τη γνώμη είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πριν από δύο εβδομάδες παρουσίασα ένα έγγραφο με την ε, Ευρωπαϊκή Πολιτική Στρατηγική για την ε, μεγαλύτερη ενεργοποίηση των μικρομεσαίων μα επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Και μάλιστα θα συζητήσω αυτό το θέμα στο Σάο Πάολο με ευρωπαίου ε, βιομηχανου που είναι εγκατεστημένοι στη Βραζιλία. Θέλω να περάσω από τα λόγια στα έργα. Θέλω να δω επιτόπου τι λειτουργεί καλά και τι, που χωλαίνει η κατάσταση ό,τι αφορά τι εξαγωγέ μα προ τη Βραζιλία για να καλύψουμε τι αδυναμίε. Γιατί πέραν των οικονομικών και πολιτιστικών μα δεσμών θα μπορούσαμε να ανανεώσουμε το διάλογό μας και την οικονομική μας ανάπτυξη. Θα σας ε, μιλήσω σύντομα για τους έξι τομείς που θέλω να προωθήσω. Καταρχήν, η δυναμική της Λατινικής Αμερικής θα πρέπει να μας ε, βοηθήσει να ενισχύσουμε την οικονομική και βιομηχανική μας συνεργασία. Όπως ξέρετε, η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να θέσει τη βιομηχανία στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της. Έχουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για να προωθήσουμε έναν ισχυρό και ανταγωνιστικό καθώς και πολύμορφο βιομηχανικό ιστό στην Ευρώπη για το 2020. Θα πρέπει να δώσουμε μια νέα όθηση στη βιομηχανική καινοτομία στην Ευρώπη, να βρούμε κατάλληλους μηχανισμούς ε, ώστε και οι ερευνητές μας και οι εργαζόμενοι μας να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους και να μπορέσουν να θέσουν τις εφευρέσει του σε εμπορία να εξυγχρονίσουμε τη βιομηχανία μα και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε το πρόσφορο έδαφο για μια υφόρη οικονομική ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόθυμη για ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων για τη βιομηχανική πολιτική με τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω ε, τον κόσμο. Και φυσικά σημαντικό εταίρο μα είναι και η Λατινική Αμερική. Δεύτερο, θέλω να ενισχύσω τη συνεργασία μα σε θέματα πολιτική μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι μικρομεσαίε επιχειρήσει διαδραματίζουν έναν αποφασιστικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα και το δυναμισμό της οικονομίας. Έχουμε 23 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη που αντιπροσωπεύουν το 99,8% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Είπα ότι είναι πολλές φορές ανεκμετάλλευτο το δυναμικό, το εμπορικό αυτό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ανάπτυξή τους και προς τα έξω, να ενισχύσουμε τις εξαγωγές τους. Νομίζω ότι με την ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής θα αξιοποιήσουμε καλύτερα το εξαγωγικό τους δυναμικό. Γιατί η ακρογωνία ως λίθος της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η νομοθετική πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, το Small Business Act στα αγγλικά. Στην Ευρώπη επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στην υποστήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας, ε, ανάπτυξης και διεθνοποίησης, δηλαδή εξόδου προς τα έξω. Νομίζω ότι μπορούμε με συντονισμένο τρόπο και ανταλλαγή απόψεων που θα έχουν τακτικό χαρακτήρα, μπορούμε να βελτιώσουμε τις πολιτικές μας. Στο εγγύς μέλλον θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε διαλόγους ε, με τους διαφόρους εταίρους μας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την καινοτομία. Τρίτο σημείο. Το σύστημα της ευρωπαϊκής προτυποποίησης ε, είναι μια αναγνωρισμένη ορισμένη διεθνώς επιτυχία και συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση μιας ενιαίας αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τη στιγμή αυτή έχουμε μια αναθεώρηση αυτής της ε, πρότασης. Το πακέτο μέτρων για την προτυποποίηση είναι τμήμα της νέας μας στρατηγικής. Και στο πλαίσιο αυτό που θα καλέσουμε κυρίως τους ε, οργανισμούς προτυποποίησης Λατινικής Αμερικής ε, για συνεργασία σε διεθνώς επίπεδο με τους δικούς μας οργανισμούς, ε, πραγματοποιούμε ένα σημαντικό βήμα. Το τέταρτο σημείο, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντικό ο ρόλο των πρώτων υλών στη διεθνή συνεργασία. Και αναφέρομαι στι βιομηχανικέ πρώτε ύλε. Δηλαδή αυτέ που δεν έχουν ούτε ενεργειακό ούτε γεωργικό χαρακτήρα. Γιατί όλοι είμαστε εξαρτημένοι από τι πρώτε ύλε και η πρόσβαση στι πρώτε ύλε αποτελεί μια κοινή πρόκληση. Ε, μια ανοιχτή και διαφανή αγορά θα πρέπει να αποτελέσει το κοινό μα στόχο και το ζητούμενο για όλου. γιατί η εξασφάλιση του ανεφοδιασμού πρώτων υλών είναι σημαντική σημαντικό θέμα για τις υγιείς οικονομικές σχέσεις. Γιατί η σπάνιση στον πρώτο υλών θα δημιουργήσει πρόβλημα σε πολλές οικονομίες και ίσως αποτελέσει και λόγο για συγκρούσεις. Εμείς είμαστε πιστός και αφοσιωμένος πελάτης της Λατινικής Αμερικής σε ό,τι αφορά τις πρώτες ύλες και μάλιστα καλό θα είναι να υπάρχει μια διαφοροποίηση της συνεργασίας Λατινικής Αμερικής και Ευρωπαϊκής ότι θα πρέπει από κοινού να έχουμε επικοδομητικό και καρποφόρο διάλογο με στόχο να υπογράψουμε και μελλοντικά συμφωνίες. Εγώ υπέγραψα μια συμφωνία με τη Χιλή πριν το καλοκαίρι. Η συνθήκη της Λισαβόνας μας επιτρέπει να διαμορφώσουμε και να αναπτύξουμε μια πολιτική τουρισμού που εμπίπτει στις δικές μου αρμοδιότητες. Ε, η παγκόσμια κατάσταση έχει αλλάξει και οι απαιτήσει των τουριστών και των καταναλωτών είναι διαφορετικές σήμερα. Έχω επίγνωση της ανάγκης να ενισχύσουμε τους θεσμούς Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής και να προωθήσουμε την αηφόρο και υπεύθυνη ανάπτυξη των τουριστικών μοντέλων. Γιατί έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για τον τουρισμό με στόχο να ενισχύσουμε τους δεσμούς της Λατινικής Αμερικής με την Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύοντας ε, τις ανταλλαγές, τουριστικές ανταλλαγές και μάλιστα σε περιόδους που δεν είναι περίοδοι εχμής για να αυξήσουμε τις τουριστικές ροές μεταξύ Ευρώπης ε, και ε, Λατινικής Αμερικής και Ρουμανίας, Ελλάδας, ε, Λιθουανίας, Πολωνίας και Χιλής, Βραζιλίας και Αργεντινής προκειμένου να έχουμε τουριστικές ανταλλαγές και στη χαμηλή περίοδο η Χιλή, η Αργεντινή και η Βραζιλία είναι οι πρώτε χώρε που επιλέξαμε γιατί εκεί έχουμε σημαντικέ ευρωπαϊκέ κοινότητε πέραν των ισχυρών οικονομικών και πολιτιστικών δεσμών. Το σχέδιο αυτό για τουριστικές ανταλλαγές θα εξυπηρετήσει όχι μόνο τις διάφορες επιχειρήσεις αλλά θα ενισχύσει του πολιτικού τους πολιτικούς μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής και μάλιστα το σχέδιο αυτό θα μπορούσαμε να το διευρύνουμε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής αν τελικά επιτυχία. Το, η συνθήκη τη Λισαβόνα αναγνωρίζει τη διαστημική πολιτική ω πολιτική αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μια συνεργασία με τη Λατινική Αμερική στο τομέα αυτό είναι απαραίτητη και μάλιστα θα συμβάλλει στην παγκόσμια προσπάθεια για μια πράσινη οικονομία που θα εναρμονίζεται στη νέα στρατηγική ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι προ το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει εμπορική, βιομηχανική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία που θα είναι ε, σημαντική σε θέματα διαστημικής ε, πλοήγησης και το, για το Γαλιλαίο που είναι το ευρωπαϊκό σύστημα GPS. Έτσι πιστεύω ότι θα μπορέσουμε με πιο φθηνό τρόπο να αντικαταστήσουμε το αμερικανικό GPS. Μάλιστα είχαμε με επιτυχία τους δύο πρώτους δορυφόρους στη Γαλλική Γουιάννα τον Οκτώβριο και θα επιταχύνουμε το χρονοδιάγραμμα της εκτόξευσης των νέων δορυφόρων ώστε ήδη από το 2014 να απολαύσουμε τις πρώτες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες ε, δορυφορικής πλοήγησης ε, έχουν σημαντική άδεια στον κόσμο και θα έχουν θετικό αντίκτυπο και για την Λατινική Αμερική σε θέματα χωροταξίας ή διαχείρισης ε, των φυσικών πόρων, της γεωργίας, ε, της εξορρυκτικής βιομηχανίας και της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Νομίζω ότι μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Παρατήρησης ε, της Γεωφυσικής Παρατήρησης, DNS, και του αντίστοιχου προγράμματος της Λατινικής Αμερικής. Έτσι θα καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές και ταυτόχρονα θα βελτιώσουμε την ε, αντιμετώπιση των θεομηνιών. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με δύο σημαντικά μήνυματα. Το πρώτο μήνυμα είναι το εξή. Μίλησα μόνο για τη Χιλή, Βραζιλία και Αργεντινή. Αλλά στόχο μου είναι να συνεργαστώ με όλε τι χώρε τη Λατινική Αμερική. Γνωρίζω ότι έχουμε εδώ ευρωβουλευτέ από πολλέ λατινοαμερικανικέ χώρε. Και γι' αυτό θα ήθελα να διατρανώσω το εξή. Ήδη είχα πρώτε επαφέ με υπουργού εξωτερικών τη Ουρουγουάη, Παραγουάη και με την υπουργό τουρισμού του Μεξικού στο Παρίσι και μάλιστα θα συσφίξω τους δεσμούς και με άλλες χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής. Το δεύτερο μήνυμα μου είναι ότι έχω υψηλές προσδοκίες από την διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής που θα λάβει χώρα στο Σαντιάγο. Άγνωστη προς το παρόν ημερομηνία. Θα ήθελα ε, οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες να με συνοδεύσουν στη διάσκεψη, αυτής, ε, στη διάσκεψη κορυφής όπως θα με συνοδεύσουν και στη Βραζιλία σε τρεις εβδομάδες. Να δημιουργηθεί ένα δίκτυο πρεσβευτών δηλαδή Λατινοαμερικάνων και Ευρωπαίων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μάλιστα όταν πήγα στη Χιλή τον περασμένο Ιούνιο υπέγραψα έξι πολιτικές συμφωνίες και θα ήθελα να τις μετατρέψω και σε νομικέ συμφωνίες και αντίστοιχε συμφωνίες να υπογράψω και με άλλε χώρε της Λατινικής Αμερικής που ενδιαφέρονται για θέματα του χαρτοφυλακίου μου. Θα ήθελα τέλος να εκφράσω την επιθυμία μου για ενισχυμένη συνεργασία και εμπορική και βιομηχανική με του εταίρους φίλους και αδερφούς μας από τη Λατινική Αμερική. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Αντώνιο Ταγιάννη. Είδατε τι άψογα ισπανικά μιλάει ο Επίτροπος και τον ευχαριστώ θερμά για την συνεχή υποστήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Eurolat. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Κολομβίας, στον κύριο Αγχελίνο Γκαρθών. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς της κολομβιανής κυβέρνησης και του κολομβιανού λαού και ιδιαίτερος του Προέδρου μας, του Χων Μανουέλ Σάντος Καλδερών. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση του Χωσέινας Ιγνάσιο Αλαφράγκα για την ε, νέα αυτή συνεδρία των Επιτροπών της Γιουρολάτ και θα ήθελα να σας μεταφέρω το μήνυμα του Προέδρου Καλδερών για την αφοσίωσή μας, την προσήλωση και την υποστήριξή μας σε αυτή την δυναμική συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Κοινοβουλίων της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Θέλουμε αυτή η δυναμική να, να μετατραπεί σε μεγαλύτερη ενότητα και διευρυμένη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Μια τέτοια ενότητα και συνεργασία θα πρέπει να στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στο σεβασμό των ελεύθερων και κυρίαρχων αποφάσεων των λαών να επιλέγουν τους ηγέτες τους με βάση τους συνταγματικούς τους κανόνες. Η Κολομβία είναι μια χώρα που προοδεύει διαρκώς και μάλιστα για 62 χρόνια ζήσαμε πραγματικά μια τραγωδία βίας, η ύπαρξη παράνομων ένοπλων, δυνάμεων, ανταρτών, παραστρατητικών δυνάμεων, εμπόρων ναρκωτικών, δημιούργησαν μεγάλο πόνο και πολλά δεινά για το λαό της Κολομβίας. Είμαστε ταυτόχρονα και μία χώρα που νομίζω ότι αξίζει να μελετηθεί. Γιατί πολλές φορές μείναμε εχμάλωτοι του πολέμου και της τραγωδίας ε, της βίας. Είμαστε μια χώρα που σήμερα βρίσκεται σε μια σημαντική οικονομική ανάπτυξη γιατί κατά Μέσο όρο έχουμε αιτήσει ανάπτυξη 5% ε, του ΑΕΠ. Είμαστε μια χώρα που ε, καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες για να μειώσουμε την εξαθλίωση, τη φτώχεια, την ανεργία. Και επίσης έχουμε επίγνωση ε, του μεγάλου χρέους που έχουμε απέναντι στο λαό μας. Η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να πηγαίνει από κοινού με την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των οικοκυριών. Ξεκινώντας από ίσω από αξιοπρεπείς μισθούς και εισοδήματα για τους εργαζόμενους μας. Και μάλιστα προσπαθώντας να καταπολεμήσουμε τις παράνομες ένοπλες οργανώσεις και να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά και την ατιμορρησία που είναι η σημαντική σύμμαχη του οργανωμένου εγκλήματος, καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες και σε θεσμικό επίπεδο για να εξασφαλίσουμε μια πολιτική σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών δικαιωμάτων, των ε, συνδικαλιστικών ελευθεριών και του περιβάλλοντος και στην προσπάθεια να καταπολεμήσουμε τις παράνομες οργανώσεις δεν ε, θυσιάσαμε κανένα θεμελιώδες δικαίωμα. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη βία, αλλά διευρύνοντας και ενισχύοντας τη δημοκρατία και δημιουργώντας ένα δρόμο για την επανόρθωση και την αποκατάσταση των θυμάτων της βίας. Είμαστε πιο ελληνικοί με τα θύματα και πιο άτεκτοι απέναντι στους δήμιους, στους ενόχους και ανοίγουμε ένα δρόμο ειρήνης, συγχώρησης και επανασυμφιλίωσης. Ο πρόεδρος Καλτερώνη είπε ότι οι πόρτε οι πύλες της ειρήνη στην Κολομβία δεν έχουν κλείσει, αλλά έθεσε και δημοσίως κάποιου όρου για το άνοιγμα αυτό των πυλών. Οι αντάρτες θα πρέπει να απελευθερώσουν όλους τους εχμαλώτους και μάλιστα χωρίς όρου. Γιατί θα πρέπει να σταματήσουν ταυτόχρονα τις πρακτικές της τρομοκρατία των απαγωγών, τη χρήση ναρκών κατά προσωπικού να απελευθερώσουν παιδιά και φίβους που στρατολόγησαν αναγκαστικά. Και το πιο σημαντικό είναι οι, οι αντάρτες Κολομβίας να τύχουν τις ίδιες αντιμετώπισης των τρομοκρατών της Ισπανίας και να αντιληφθούν ότι αυτό που επιθυμεί ο λαός μας είναι να ζει εν ειρήνη και χωρίς βία. Μάλιστα, σήμερα έχουμε αναπτύξει και ένα πρόγραμμα διεθνούς συνεργασίας συνεννόησης ε, με όλες τις χώρες του κόσμου, ξεκινώντας φυσικά από τις γειτονικέ μας χώρες. Αποδίδουμε ιδιαίτερα σημασία στην ε, ενότητα στην περιοχή μας. Ε, θέλουμε να δώσουμε έμφαση στους μηχανισμούς ολοκλήρωσης και θα δείξουμε σεβασμό στις απόψεις ε, των κυβερνήσεων και των λαών των γειτονικών χωρών. Και από αυτή την άποψη θα θέλαμε η συνεδρία αυτή της Eurolat να λάβει υπόψη και την κατεύθυνση που θα λάβουν οι συμφωνίες σύνδεσης, οι εμπορικές συμφωνίες, οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και στην περίπτωση της Κολομβίας θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για τις συνεχείς προσπάθειές μας και την αδιάκοπη συνεργασία μας με όλες τις χώρες του κόσμου, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Ιαπωνία, την Κίνα, την Νότιο Κορέα, με τις χώρες της περιοχής και φυσικά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος μας είναι να υπογράψουμε εμπορικές συμφωνίες και στα πλαίσια των εμπορικών συμφωνιών προσπαθούμε να εφαρμόσουμε και τη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, ε, τα εργασιακά δικαιώματα και το σεβασμό του περιβάλλοντος. Τέλος, ήθελα να πω ότι πιστεύω πως όλοι οι πολυμερείς οργανισμοί, αλλά και οι περιφερειακές οργανώσεις, θα έπρεπε να συζητήσουν εμβριθώς και διεξοδικά πώς στα πλαίσια των εμπορικών συμφωνιών θα σημειώσουν πρόοδο και για συμφωνίες που θα σέβονται πλήρω τα ανθρώπινα δικαιώματα. Χρειαζόμαστε εμπορικέ συμφωνίε που θα έχουν όμω ανθρώπινο πρόσωπο. Θέλουμε εμπορικέ ε, συμφωνίε που θα θέσουν στο επίκεντρό τους το σεβασμό και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, ξεκινώντας από τα παιδιά. Σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στην Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Κολομβίας βρισκόμαστε στη φάση της κύρωσης ε, της συμφωνίας αυτής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κολοβιανή Βουλή. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι εδώ δεν ζητούμε χάρες, ούτε θέλουμε να κάνουμε χάρες. Δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει εδώ χάρη στην Κολομβία, ούτε η Κολομβία κάνει καμιά χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε η εμπορική αυτή συμφωνία να ευνοήσει την οικονομική ανάπτυξη και τις πολιτικές απασχόλησης και, στις, και στους διαιτέρους. Θα πρέπει και οι δύο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κολομβία να βγουν κερδισμένοι από την εμπορική συμφωνία. Από κοινού θα δημιουργήσουμε ένα μέτωπο για να μεριμνήσουμε για την πλήρη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και στα πλαίσια αυτής της εμπορικής συμφωνίας που ε, θα ακυρώσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, θα πρέπει να δούμε πώς γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα εδώ, αλλά και η κολομβιανή κυβέρνηση, η κολομβιανή βουλή και ο κολομβιανός λαός θα μεριμνήσουν για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κολομβία. Για μας σημαντικό είναι οι σχέσεις, οι αμοιβέ σχέσεις μας να μην περιοριστούν μόνο σε εμπορικές συμφωνίες. Το πιο σημαντικό για μας είναι η ταυτότητα των αξιών, των δημοκρατικών αξιών. Και τμήμα αυτής της ταυτότητας των δημοκρατικών αξιών έγκυται στο γεγονός ότι στα σύγχρονα κράτη ο βασικός άξονας είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, το δικαίωμα ελεύθερη έκφραση, η ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών. Αυτοί είναι οι άξονες των δημοκρατικών μας αξιών. Και μια άλλη σκέψη που θα μπορούσαμε να κάνουμε στο πλαίσιο της Eurolat είναι ακριβώς αυτή, γιατί κατά τη γνώμη της Κολομβίας η δυναμική της παγκοσμιοποίησης των εμπορικών συναλλαγών, της εμπορικής παγκοσμιοποίησης, αυτή η δυναμική είναι αναπόφευκτη. Και θα πρέπει στη δυναμική αυτή, στις πολυμερείς οργανώσεις, να βρούμε μηχανισμούς ώστε να συμπεριλάβουν στις εμπορικές συμφωνίες και τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την πολιτική ακριβοδίκαιων μισθών και αμοιβών. Όπως είπαμε σε πολλές περιπτώσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και στην Λατινική Αμερική, η Κολομβία για παράδειγμα, μαστίζονται από εσωτερική βία, από διάφορες δράσεις οργανωμένου εγκλήματος, ταλανίζονται από την ύπαρξη παράνομων ε, ενόπλων οργανώσεων. Μερικές χώρες ζούμε τις συνέπειες της τρομοκρατίας, βιώνουμε τις συνέπειες του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, του παράνομου εμπορίου όπλων, της σωματεμπορίας και έχουμε την εντύπωση ότι φέρουμε την υποχρέωση, φέρουμε την ευθύνη να βρούμε τρόπους συνεργασίας μεταξύ των διαφορών χωρών. Γιατί μιλούμε για διασυνοριακά εγκλήματα. Για εγκλήματα που δεν περιορίζονται, δεν σέβονται σύνορα. Και τα εγκλήματα αυτά, αν δεν τα αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα, θα θα μπορούσαν να κλονίσουν τη δημοκρατία ή τους δημοκρατικούς θεσμούς σε οποιαδήποτε χώρα. Τα εγκλήματα αυτά στηρίζονται στην διαφθορά και στην ατιμορρησία. Ουσιαστικά υπονομεύουν δηλαδή και το δικαστικό μηχανισμό και το μηχανισμό απονομής δικαιοσύνης. Σήμερα η Κολομβία έχει στο πρόγραμμά της το διάλογο και τη συνεργασία με πάνω από 40 χώρες του κόσμου. Και στην προσπάθεια, στην προσπάθεια αυτή έχει συμπεριλάβει και την καταπολέμηση των εγκλημάτων. Βασικό άξονα τη συνεργασία μας με τις άλλες χώρες δεν είναι κάποια ιδεολογικά κριτήρια ή ιδεολογική συνάφεια με τις διάφορες κυβερνήσει και τους κυβερνώντες. Ο κοινό μα άξονα είναι ότι οτιδήποτε παράνομο αντίκειται στη δημοκρατία. Ότι οτιδήποτε παράνομο συνομωτεί κατά τη δημοκρατία. Οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, είτε ε, είναι διαφθορά, είτε ατιμορρησία, είτε οργανωμένο έγκλημα, συνομωτεί ε, κατά της ευημερία και του δικαιώματος των πολιτών να ζουν ε, σε ηρεμία και ειρήνη. Έχουμε την αίσθηση ότι αυτή η συνεδρίαση της Γιουρολάτ θα μπορούσε να μας βοηθήσει ώστε να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς συνεργασίας, της διμερούς ή της πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών για να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα, τη βία, να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία, το λαθρεβόριο των ναρκωτικών και οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα. Ταυτόχρονα έχουμε την αίσθηση ότι μας παρουσιάζεται μια καταπληκτική ευκαιρία, μια μοναδική ευκαιρία στο πλαίσιο των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής, μια μοναδική ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων, πρακτικών, για να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε την κρίση αυτή. Εμείς στην Κολομβία είμαστε αισιόδοξοι. Αισιοδοξούμε ότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με όλη αυτή την παράδοση της ολοκλήρωσης, της συνεργασίας, του αγώνα για τη δημοκρατία και την ειρήνη που έχει η Ευρώπη, οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών, τα κοινοβούλια, τα κόμματα και η κοινωνία των πολιτών θα καταφέρουν να βρουν λύσεις για διέξοδο από την κρίση. Την κρίση που μαστίζει ιδιαίτερα ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιθυμία της δικής μας κυβέρνησης είναι αυτή και το εκδηλώσαμε αυτό σε πολλές περιπτώσεις. Πιστεύουμε και αισιοδοξούμε ότι θα ε, βγούμε από την κρίση. Γιατί έχουμε επίγνωση ότι αυτή η κρίση μπορεί να επηρεάσει και εμάς. Θα ήθελα επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί με μεγαλύτερη ηρεμία και νυφαλιότητα να αναλύσει τις εμπειρίες, τις διάφορες εμπειρίες των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Και το τι έκαναν αυτές οι χώρες για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης του 2008. Μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που δεν τη δημιουργήσαμε εμείς. Μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που τη δημιούργησε και την προκάλεσαν άλλοι. Εμείς στη Λατινική Αμερική καταφέραμε με σχετική επιτυχία να εξέλθουμε από την κρίση. Δεν είμαστε βέβαια πλήρως προστατευμένοι, ούτε είμαστε θωρακισμένοι, αλλά νομίζω ότι σημειώσαμε πρόοδο, μεγαλύτερη ή μικρότερη, σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης, σε θέματα ενίσχυσης της απασχόλησης. Και αυτό το δρόμο συνεχίζουμε να ακολουθούμε στην Ευρω... στη Λατινική Αμερική. Και στην κατεύθυνση αυτή Δώσαμε ιδιαίτερο στόχο στην ενότητα, στη συνεργασία. Συγκαλέσαμε ε, συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών των χωρών της περιοχής για να δούμε τι άλλες πρωτοβουλίες μπορούμε να αναλάβουμε. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε το διάλογο μεταξύ εργαζομένων, εργοδοτών και κυβερνήσεων για να αποτρέψουμε τις συνέπειες μιας νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Και πιστεύω ότι σήμερα η Λατινική Αμερική, η περιοχή μας, η Λατινική Αμερική των κυβερνήσεων των ιδιωτεροτήτων είναι μια περιοχή που με τις εμπειρίες της να δείξει ότι ενωμένη μπορούμε να επιλύσουμε και τα εσωτερικά μας προβλήματα. Θα ήθελα να ολοκληρώσω εδώ επαναλαμβάνοντας και διατρανώνοντας τη βούληση της κυβέρνησης ε, της Κολομβίας αλλά και της ε, κοινωνίας της Κολομβίας να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ε, συνεργασίας και της ενότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής. Αυτό είναι ο δικός χάρτης για μας, αυτή θα είναι η πορεία μας και ως εκ τούτου τα συμπεράσματα αυτής της εκδήλωσης όχι μόνο θα τα λάβουμε υπόψη στα κοινοβούλια μας, αλλά να είστε βεβαίοι ότι και η Κολομβιανή κυβέρνηση θα λάβει τα συμπεράσματα αυτά ως σημείο αναφοράς για τις διάφορες πολιτικές της, που στόχο έχουν τον καθημερινό αγώνα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των Κολομβιανών πολιτών, εν ειρήνη και εν ηρεμία. Γιατί η διακυβέρνηση έχει νόημα, όπως και η δημοκρατία έχει νόημα, όταν φέρει στο επίκεντρό τη τα ανθρώπινα όντα και κυρίως τα παιδιά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε της Δημοκρατίας Κολομβίας, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και για την ε, αδιάλειπτη υποστήριξή σας στις εργασίες της Eurolat. Το λόγο έχει τώρα η πρόεδρος του Ιδρύματος Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής, η κυρία Μπενίτα Φερέρο Βάλτερ. Σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ καταρχήν θερμά τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, την κυρία Οκέλη και τον κύριο Σαλαφράγκα, τον Αντιπρόεδρο Ταγιάννη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να τον ευχαριστήσω την Γενική Γραμματέα της Ουνασούρ, τον Αντιπρόεδρο της Κολομβίας, τη Γενική Γραμματέα της ΕΠΑΛ, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, εξοχότατοι. Θα ήθελα να εκφράσω την ε, μεγάλη χαρά που αισθάνομαι για τη συμμετοχή μου σε αυτή την πανηγυρική συνεδρίαση της συνέλευσης της Eurolat. Ανέλαβα ε, πρόσφατα την Προεδρία του Ιδρύματος EU-LAC και με βάση τη νέα μου ιδιότητα, είναι η πρώτη φορά που εμφανίζομαι εδώ στην Σύνοδο της Γιουρολάτ από τότε που ολοκληρώθηκε η θητεία μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην πρώτη επιτροπή του Χωζέ Μανώλη Μπαρόζο. Πριν από πέντε χρόνια, στις, ε, στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής ε, που έγινε στη Βιέννη, συμμετείχα στην κατάρτιση μιας πρότασης που τότε ήταν ένα όραμα, ένα όνειρο και σήμερα έγινε πραγματικότητα, έλαβε σάρκα και οστά. Και αυτό το όνειρο ήταν η ίδρυση του Ιδρύματος Ευρωπαϊκής Ένωση και Λατινική Αμερική Καραϊβικής. Γιατί τότε προβληματιζόμασταν ποιο θα μπορούσε να είναι ο ρόλος της κοινωνία των πολιτών και στις δύο περιοχές. Και όταν λέγαμε κοινωνία των πολιτών, εννοούσαμε την κοινωνία των πολιτών με ευρία έννοια. Είχαμε τότε αντιληφθεί ότι η στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο περιοχών που ήδη υπήρχε σε κυβερνητικό επίπεδο θα έπρεπε να τύχει κάποιες εμβάθυνσεις και ενίσχυσης και σε άλλα επίπεδα. Εξού και η ιδέα μας να ιδρύσουμε ε, ένα ίδρυμα, μία απόφαση που έλαβε η ε, Σύνοδος Κορυφής της Μαδρίτης πέρυσι το Μάιο, το Μάιο του 2010. Θα ήθελα στα συμπεράσματα της Μαδρίτης να αναφερθώ, γιατί εκεί προσδιορίζονται ε, προσδιορίζεται ο στόχος της Γιουρολάτη. να γίνει ένα σημαντικό, ένα χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας και να δώσει τροφή για τη συζήτηση για τις κοινέ στρατηγικές και δράσεις προκειμένου να ε, βελτιωθεί η προβολή αυτού του Ιδρύματος. Τελικά έγινε η ίδρυσή του και εγγενιάστηκε στις 7 Νοεμβρίου στο Αυγούργο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον ε, συμπρόεδρο που βρέθηκε εκεί. Είχαμε, ε, συνήψαμε πολλές συμφωνίες με στρατηγικούς εταίρους. Μία στη, στο Παρίσι, τη Γαλλία και στη, στο Μιλάνο της Ιταλίας. Ευελπιστώ ότι και οι φίλοι μας της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής θα έχουν προνομιούχους ε, εταίρους με παρόμοιους όρους ε, που έχουμε και εμείς. Φυσικά από εσά εξαρτάται ποιοι θα είναι οι εταίροι σας, οι προνομιακοί αυτοί εταίροι. Η ε, Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής ήταν ανέκαθεν σημαντικός φορέας προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των δύο υπήρων. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Eurolat, τον Χωσέ Γνάσιο Αλαφράγκα, αλλά και όλους εσάς για την αδιάλειπτη υποστήριξή σας στις σχέσεις ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής Καραϊβικής και ιδιαίτερα για τη συμβολή σας στην ίδρυση αυτού του νέου οργανισμού, του νέου ιδρύματος. Και ευελπιστώ ότι θα συνεχιστεί αυτή η αμέριστη υποστήριξή σας για να ανταπεξέλθουμε στο τεράστιο έργο μας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω φυσικά και για τη σημερινή πρόσκληση. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βέβαια ο Αντιπρόεδρος έφυγε, έδειξε από την αρχή μία αφοσίωση και μία υποστήριξη προς το Ίδρυμα αυτό που χρήζει ειδική μνήμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και προσωπικά τον πρόεδρο Μπαρόζο για την πολύ επικοδομητική του συμβολή, αλλά και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, καθώς και όλους τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το άοκνο έργο που επιτέλεσαν ε, όλο αυτό τον καιρό για το Ίδρυμα Ιούλακ. Και θα ήθελα να πω στον Αντιπρόεδρο Ταγιάννη ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας είπε, γιατί εστερνιζόμαστε πολλά από αυτά που μας είπε, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τη συνεργασία σε πολλούς τομείς. Και εμείς, το Ίδρυμά μας, θα διαδραματίσει ρόλο πλατφόρμας για την ενίσχυση αυτής της συνεργασίας. Και εκ μέρους του εκτελεστικού διευθυντή που είναι παρόν και εκ μέρους του πρέσβη Χόρχε Βαλδές, αλλά και ε, προσωπικά να σας ευχαριστήσω θερμά και μέσω ημών να ευχαριστήσω όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Καραϊβικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκριση του καταστατικού του Ιδρύματος EU-LAC. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη γερμανική κυβέρνηση που διευκόλυνε την σύσταση αυτού του Ιδρύματος. Γιατί η αρχή ήταν δύσκολη και τελικά η πόλη του Αμβούργου έδειξε την προθυμία της ε, και τη συνεργασία της. Και νομίζω ότι η επιλογή ήταν πολύ θετική και θα έχουμε στενή συνεργασία και με το Δήμο του Αμβούργου. Κυρίες και κύριοι, στις πρόσφατες επισκέψεις που έκανα στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, αντιλήθηκα τις υψηλές προσδοκίες που έχουν οι χώρες αυτές από το Ίδρυμά μας, από το Νεοπαγές αυτό Ίδρυμα, ιδιαίτερα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έχουμε τεράστιες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και γι' αυτό θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την συγκυρία που χθε η Αλήσια Μπάρσανα τη χαρακτήρισε ως σημείο καμπής που θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Εγώ θα έλεγα όχι μόνο σημείο καμπής, θα έλεγα και σημείο ε, εμβάθυνσης για τις υπάρχουσες σχέσεις που όμως έχουν και ένα αναξιοποιητό μέχρι στιγμής δυναμικό. Έχω επίγνωση ε, της πληθώρας των θεσμικών οργάνων και των οργανώσεων που υπάρχουν για την προώθηση των σχέσεων μεταξύ των δύο υπήρων. Παρ' όλα αυτά το δικό μας Ίδρυμα, το Ίδρυμα EU-LAC, Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής, είναι το μοναδικό Ίδρυμα στο οποίο συμμετέχουν και οι 60 χώρες που απαρτίζουν αυτή τη στρατηγική συμμαχία. 27 και σύντομα 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι 33 χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Όλες αυτές οι χώρες συμμετέχουν σε μια κοινή πλατφόρμα, το Ίδρυμα e ULAC. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα ε, ε, να σας πω δύο λόγια για το αντικείμενο του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα EuroLac έχει στο αντικείμενο να ενθαρρύνει την αμοιβαία γνώση και κατανόηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής καθώς και περιοχών της Καραϊβική και των λαών αυτών των περιοχών. Είναι ένα ευρύ στόχο, είναι ευρύ αντικείμενο, αλλά είναι σαφή ο στόχο όλων. Η κοινωνία των πολιτών είναι στο κέντρο αυτών που κάνουμε και ο βασικό μα στόχο θα είναι να ενισχύσουμε και να εμβαθύνουμε με τη συνεργασία μεταξύ των δύο περιοχών να βελτιώσουμε τις ε, διαπολιτισμικές συνεργασίες και τη γνώση και τη φιλία μεταξύ των λαών μας μέσω ε, της συνεισφοράς της κοινωνίας των πολιτών ε, και άλλων κοινωνικών φορέων. Θέλουμε η κοινωνία των πολιτών να είναι το βασικό στοιχείο του Ιδρύματός μας. Είναι σημαντικό διότι ε, είμαστε πεπισμένοι από τα πλεονεκτήματα τα οποία θα έχουν όλοι οι συμβαλόμενοι από αυτό και παράλληλα διότι η κοινωνία των πολιτών πρέπει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες που προσφέρουν και οι δύο περιφέρειές μας, ούτως ώστε η κοινωνία των πολιτών να μπορέσει να συμμετέχει και να υποφελείται από αυτή τη στρατηγική σχέση. Γι' αυτό τον λόγο είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη που ακούω ότι ο Αντιπρόεδρος Ταγιάννη έχει την πρόθεση να υποστηρίξει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θέλει να δουλέψει και στον τομέα του τουρισμού και έχει και πολλές άλλες πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες που θα ενισχύσουν και την βιομηχανία αλλά τελικά όπως είπε χθε η Αλήθεια Μπάρθενα θα βελτιώσει και την ευημερία των πολιτών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κυρίες και κύριοι, θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το Ίδρυμα ώστε να γίνει σημείο αναφοράς ενός δικτύου συνεργασίας και συντονισμού που όλοι θα συντονίζουμε τις προσπάθειές μας, αναγνωρίζοντας φυσικά τις ε, διάφορες οργανώσεις και το ρόλο τους ε, συνεργασίας ε, της κυβέρνησης και της κοινωνίας των πολιτών. Ο πυρήνας του Ιδρύματος θα είναι οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρηματίες, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκπρόσωποι συνδικαλιστών, βουλευτές, εσείς, άλλα ιδρύματα, πανεπιστήμια, ε, πανεπιστημιακοί κύκλοι, κέντρα ανάλυσης, μη κυβερνητικέ οργανώσεις και ούτω καθεξής. Θα θέλαμε η κοινωνία των πολιτών να αντιληφθεί όλες αυτές τις δυνατότητες που υπάρχουν και να τις αξιοποιήσει. Θέλουμε να γίνουμε ένα υπόδειγμα και σημείο αναφοράς για την πρόθεση των ανταλλαγών. Πρώτα απ' όλα όμως θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι, θέλουμε να βοηθήσουμε. Το Ίδρυμά μας, κατά τη γνώμη μου, βρίσκεται σε προνομιούχο θέση και μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών μεταξύ των διαφόρων μελών του. Μέχρι στιγμή η δράση ήταν παράλληλη όλων αυτών των φορέων. Χάρη στο Ίδρυμα σήμερα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε διασταυρωμένες ε, ε, σχέσεις, ε, εγκάρσεις, πολυμερείς και να μην είναι πια παράλληλοι δρόμοι. Βέβαια έχουμε μπροστά μας πολύ μακρύ δρόμο να είναι πραγματικά αποδοτικό αυτό το Ίδρυμα και χρήσιμο. Κάναμε τα πρώτα βήματα που είναι πολύ σημαντικά, αλλά δεν θα πρέπει να περιοριστούμε σε αυτή την πρόοδο. Βρεθήκαμε στην πρώτη φάση της συγκρότησης του Ιδρύματος, εγκρίναμε τα καταστατικά με βάση ε, το Γερμανικό Σύνταγμα και η έδρα μας βρίσκεται στο Αμβούργο. Στη δεύτερη φάση τώρα, στόχος μας είναι να γίνουμε ένας πραγματικά διεθνής οργανισμός, μια διεθνής οργάνωση. Και αυτός ε, ο νομικός χαρακτήρας θα μας επιτρέψει, ε, αυτή η νομική προσωπικότητα θα μας επιτρέψει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη διεκπαιρέωση του στόχου μας, του των στόχων μας. Έτσι θα μπορέσουν και οι 60 χώρες μέλη του Ιδρύματος να συμβάλλουν πλήρως ε, στη λειτουργία του Ιδρύματος αλλά και στη χρηματοδότησή του που είναι και αυτή απαραίτητη. Κυρίες και κύριοι, έχω σημειώσει πολλά εδώ πέρα στην ομιλία μου αλλά βλέπω ότι ο χρόνος προχωρεί, δεν θα ήθελα να σας κουράσω. Θα ήθελα απλώς να πω ότι οι στόχοι και το περιεχόμενο του Ιδρύματος θα καλύψουν όλα τα θέματα των διασκέψεων κορυφής Κατά πολέμηση της ε, φτώχειας, θέματα παιδείας, ε, κατάρτισης, απασχολησιμότητας, φορολογικές, δημοσιονομικές πολιτικές, καταπολέμηση τρομοκρατίας, ε, λαθρεμπορίων ναρκωτικών, κλιματικές αλλαγές, ασφάλεια του πολίτη, χρηστή διακυβέρνηση και φυσικά εμπέδωση της δημοκρατίας. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και ένα πρόγραμμα δράσεων της Μαδρίτης, δηλαδή τα νέα θέματα, την έρευνα, την καινοτομία, την τεχνολογία και τώρα για την επόμενη διάσκεψη κορυφής του Σαντιάγο της Χιλής, ε, χιλή, ε, με περιβαλλοντικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε μπροστά σε μια ε, ιστορική ευκαιρία. Οι πολιτικές, θεσμικές και οικονομικές μας σχέσεις έχουν ήδη φτάσει σε ένα βαθμό ρημότητας που θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε, να βελτιώσουμε, να εμπεδώσουμε ε, μία πιο ορατή πια σχέση που θα φτάσει και θα αγγίξει όλους τους πολίτες μας. Πιστεύω ότι το Ίδρυμά μας θα έχει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που θα συμβάλλει και θα βοηθήσει τους πάντες. Και με τη σύσταση αυτού του Ιδρύματος ε, εσαρκώνουμε το όνειρο που ήταν κοινό όνειρο όλων μα που δώσαμε ραντεβού εδώ σήμερα. Θα ήθελα να σα πω ότι ο εκτελεστικό διευθυντής και ο πρέσβη Χόρχε Βαλντέ και εγώ ω πρόεδρο του ιδρύματο αυτού προσβλέπουμε σε συνεργασία μαζί σα και υπολογίζουμε στην υποστήριξη και τον ενθουσιασμό σα. Κυρίω στον ενθουσιασμό των Ευρωβουλευτών αλλά και των μελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Eurolat έχω την ακράδαντη και ειλικρινή πεποίθηση ότι αυτό το σχέδιο αξίζει και τις προσπάθειες και την εκτίμησή μας. Γιατί αντιμετωπίζουμε μία μοναδική ευκαιρία. Δεν μπορούμε να χάσουμε αυτό το τρένο, δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε του Ιδρύματος EULAC να είστε βεβαία ότι όλη η υποστήριξη που μας είχατε προσφέρει τότε ως Επίτροπος για να προωθήσουμε τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής θα σας την ανταποδώσουμε ακόμη πιο ενισχυμένη στο έργο σας ως Πρόεδρο του Ιδρύματος. Θα δώσω τώρα το λόγο στην ε, εκτελεστική γραμματέα της ε, ΕΚΛΑΚ, της Οικονομικής Επιτροπής Λατινικής Αμερικής και ε, Καραϊβικής, την κυρία Ελίσια Μπάρσενα. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Θα ήθελα με ιδιαίτερη στοργή και εκτίμηση να απευθύνω θερμό χαιρετισμό προς τον κύριο Σαλαφρά και να τον ευχαριστήσω για την πρόσκληση συμμετοχή στη Eurolat. Θα ήθελα να χαιρετήσω την Μπερνίτα Φερέρο, τον Χόρχε Μπαλδές, την αγαπητή φίλη Μαρία Εμαμεχία, τον Δον Αγχελίνο Γκαρσόν, τον σύντροφο, την Κλάουρια Ορκέλη, και όλους εσάς ε, φίλες και φίλους και κυρίως τους βουλευτές της Λατινικής Αμερικής και να σας πω ότι αυτή είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική ευκαιρία και λαμβάνει η χώρα μια στιγμή τεράστιων αλλαγών, σε ένα σημείο καμπή. Γιατί πραγματικά σε αυτό το σημείο καμπή βρίσκεται ο κόσμο σήμερα και δημιουργείται ένα νέο σενάριο με τους πολίτες που συμμετέχουν πιο έντονα, είναι καλύτερα κατατοπισμένοι και απαιτούν ε, ε, πληροφόρηση για τις εξελίξεις και απαιτούν από εμά, αλλά κυρίως από εσά, τους βουλευτές, εξηγήσει. Οι πολίτες ζητούν από όλους τους πολιτικούς εξηγήσει ε, για το πώς σκοπεύουμε να διαμορφώσουμε τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής, γιατί τα πράγματα θα αλλάξουν. Όπως είπε και ο Επίτροπος, ο Τον Αντώνιο Ταγιάννη, και η Ευρώπη θα βγει διαφορετική από την κρίση, αλλά και η Λατινική Αμερική είναι ήδη διαφορετική. Θα πρέπει να βρούμε ένα νέο τρόπο για να εστιάσουμε τη συνεργασία μας με νέο όραμα που θα συνδυάζει την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και πρώτα απ' όλα κοινωνική ένταξη και συμμετοχή. Αυτό προϋποθέτει πολιτικές ε, που στόχο θα έχουν την αντιμετώπιση των βασικών ανισοτήτων των, ε, της Λατινικής Αμερικής. Γιατί η Λατινική Αμερική δεν είναι η φτωχότερη ήπειρος του κόσμου, αλλά η ήπειρος με τις μεγαλύτερες ανισότητες, το είπαμε. Και ε, η Ουρουάη που έχει το καλύτερο ΑΕΠ της περιοχής και τις λιγότερες ανισότητες έχει αντίστοιχο ΑΕΠ με τις Φιλιππίνες που είναι η, πιο, η χώρα με τις μεγαλύτερες ανισότητες της Ασίας για να σας δώσω ένα μέτρο σύγκρισης. Έχουμε λοιπόν τεράστιες προκλήσεις και σήμερα αντιμετωπίζουμε και μεγάλη αβεβαιότητα. Μία αβεβαιότητα με τουλάχιστον δύο ταχύτητες ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Υπάρχει μία στασιμότητα στις ε, ανεπτυγμένες βιομηχανικές χώρες και μία ε, επιβράδυνση ακόμη και στις αναπτυσσόμενες χώρες, αν υπάρχει μία επιτάχυση σε κάποιες αναδυόμενες οικονομίες. Η παρούσα οικονομική κρίση στην Ευρώπη, θα, αντί να μας απομακρύνει, θα πρέπει να μας φέρει πιο κοντά. Θα πρέπει να μας φέρει πιο κοντά ακριβώς γιατί δημιουργεί ένα παράθυρο ευκαιρίας για να δώσουμε ένα νέο δυναμισμό σε αυτή τη διαπεριφερειακή συνεργασία και να την εφοδιάσουμε μια νέα οπτική και ένα νέο βλέμμα. Εμείς στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική αντιμετωπίζουμε τη συγκυρία αυτή με πολύ σημαντικά εφόδια που συγκεντρώσαμε τις τελευταίες δεκαετίες. Από τη μία πλευρά έχουμε μια εμπέδωση της δημοκρατίας και των δημοκρατικών θεσμών. Παρά τις δυσκολίες έχουμε πια μια περιοχή που είναι κατεξοχήν δημοκρατική με μια ανάπτυξη σταθερή με εξαίρεση το 2009 και δημιουργήσαμε μια μακροοικονομική ανάπτυξη και έχουμε μακροοικονομικού δεσμού. εφαρμόζουμε μια μακροοικονομική προνοητικότητα, όπω δείχνουν οι δείκτες. Σήμερα το εξωτερικό χρέο, για παράδειγμα το δημόσιο χρέο στη Λατινική Αμερική είναι τη τάξη του 30% του ΕΠ. Έχουμε διεθνή αποθέματα άνω των 750 δισεκατομμύριων δολαρίων και ίσως το πρόβλημα, το πιο σημαντικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε στο εγγύς μέλλον ε, θα είναι το έλλειμμα του τρέχοντος λογαριασμού. Και αυτή είναι η διαφορά με την κρίση του 2008 που οι περισσότερες οικονομίες μας είχαν πλεόνασμα τέτοιο εμπορικό. Κάτι που μας δημιουργεί πιο στενό δημοσιονομικό πλαίσιο για να αναλάβουμε μέτρα κατά της κρίσης. Περάσαμε από μια περίοδο δυναμισμού, όπως είπαμε, στη Λατινική Αμερική. Είχαμε ανάπτυξη το 2010 μέχρι και 6%. Φέτος ε, θα έχουμε 4,4% οικονομική ανάπτυξη, το 2012 3,8%. Υπάρχει μια επιβράδυνση δηλαδή. Βλέπετε ότι υπάρχει μια μικρή επιβράδυνση, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική ε, είναι ε, ανθεκτικές απέναντι στις εξωτερικές διαταραχές και αυτό χάρη στις δύο δεκαετίες που εφαρμόσαμε οικονομικές μεταρρυθμίσεις, που εμπεδώσαμε τους θεσμούς και εφαρμόσαμε μεγαλύτερη προνετικότητα δημοσιονομική και νομισματική. Και επίσης έχουμε και αυστηρότερη νομισματική επιτήρηση. Έχουμε όμως και το θέμα, της, το θέμα, το θέμα των τραπεζών στη Λατινική Αμερική. Και μάλιστα για να ενισχύσουμε την οικονομική ανάπτυξη, θέλουμε μεγαλύτερη τραπεζική πυκνότητα. Εκεί είναι που χωλαίνει η κατάσταση στη Λατινική Αμερική. Άλλο πολύ σημαντικό είναι ε, ότι στη Λατινική Αμερική καταφέραμε τα τελευταία 20 χρόνια να μειώσουμε τη φτώχεια αισθητά. Και μεταξύ της δεκαετίας του 1990 και του 2010 πραγματικά κατορθώσαμε να μειώσουμε την φτώχεια κατά 12% και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξεκινήσαμε ε, με τη χαμένη δεκαετία του 80 με τους μισούς Λατινοαμερικανούς να είναι φτωχοί και σήμερα ε, το ποσοστό των φτωχών είναι 32%. Δεν μιλάμε για μελιτέο ε, ποσό, μιλάμε για 180 εκατομμύρια Λατινοαμερικανών που είναι φτωχοί και 66 εκατομμύρια βρίσκονται σε κατάσταση εξαθλίωσης. Έχουμε τεράστιο έργο μπροστά μας για να δημιουργήσουμε πιο ίσες, ισότιμες κοινωνίες. Βελτιώσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία της περιοχής ε, μείωση των ανισοτήτων στο δίκτυο του Gini και έχουμε ανεργία 7,3%. Βέβαια, έχουμε κάποια αριθμητικά στοιχεία που ε, κρύβουν μια τραγική κατάσταση στη Λατινική Αμερική που είναι ο άτυπος χαρακτήρας, οι μη δηλωμένε θέσει εργασία. Βέβαια είχαμε 12 εκατομμύρια Λατινοαμερικάνους που μπήκαν στη μέση τάξη τα τελευταία χρόνια και υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες οικονομικής ανάπτυξης. Αλλά υπάρχουν και περισσότερες απαιτήσει από τις κυβερνήσεις, από το δημόσιο τομέα για ποιοτικές κοινοφελείς υπηρεσίες όπως είναι η παιδεία, για παράδειγμα. Και γι' αυτό και η Λατινική Αμερική γίνεται όλο και πιο ελκυστική αγορά και για τους εξαγωγείς και για τους επενδυτές. Όπως πολύ σωστά μας είπε ο ε, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Αντώνη Ταγιάννη, έχουμε και πλούσιο ρηκτό πλούτο. Ξάγουμε το 42% του χαλκού του κόσμου, 47% της σόγιας παγκοσμίω. Είμαστε μια περιοχή με πολλούς προ... πολλές πρωτεσίλες, είμαστε σιτοβολώνας και φυσικά έχουμε και ένα τρίτο της, των αρδεύσιμων καλλιεργιών, ένα τρίτο του νερού, 30% ε, των δασών παγκοσμίω. Έχουμε πάρα πολλές πρώτες αλλά έχουμε και ένα κόδωνα του κινδύνου. Να επανέλθει η οικονομία στον πρωτογενή τομέα Δηλαδή, εγκυμονεί ο κίνδυνο να μην καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε προστιθέμενη αξία στα αγαθά και τι υπηρεσίε, τουλάχιστον στα αγαθά που εξάγουμε εμεί. Και εκεί έγκυται η σημαντική πρόκληση για μα. Γι' αυτό και ευελπιστούμε ότι σε αυτό το νέο στάδιο των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα πραγματοποιούμε μια ανάλυση που ελπίζω ότι θα την κάνουμε από κοινού πριν την επόμενη διάσκεψη κορυφής, για τις επενδύσεις. Μία ανάλυση για τις επενδύσεις. Γιατί πολλοί λένε ότι η Κίνα θα γίνει ο νέος γίγαντας που θα έρθει για επενδύσει στη Λατινική Αμερική. Ήδη η Κίνα είναι παρούσα στη Λατινική Αμερική. Και φυσικά η παρουσία της γίνεται όλο και πιο αισθητή εκεί. Γίνεται ατμομηχανή η Κίνα για την οικονομία παγκοσμίω. Οι ευρωπαϊκέ επενδύσει όμω που έφτασαν στη Λατινική Αμερική, καταρχήν δεν είναι μόνο ισπανικέ και πορτογαλικέ αυτέ οι επενδύσει. Χθε το συζητούσαμε αυτό όλη τη μέρα. Οι ευρωπαϊκέ επενδύσει έχουν σημαντική διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά την προέλευση του ε, και του τομεί. Και μάλιστα οι ευρωπαϊκέ επενδύσει είναι παρούσες στη Λατινική Αμερική δεκαετίες ολόκληρε σε μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων και περισσότερο δραστηριοτήτων βιομηχανικών, μεταποιητικών παρά εξορρυκτικών δραστηριοτήτων. Και χάρη σε αυτές τις επενδύσεις βελτιώνουμε τις προδιαγραφές μας σε ό,τι αφορά την προστασία των εργατικών δικαιωμάτων, ε, ευαισθητοποιούμαστε περισσότερο για το περιβάλλον και έχουμε τέτοιες επενδύσεις που δημιουργούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης και ε, προβαίνουν και σε μια μεταφορά τεχνολογίας. Υπάρχει και τεχνολογική πρόοδος λοιπόν χάρη σε αυτέ τι ευρωπαϊκέ επενδύσει. Και αυτό προσπαθούμε να το εξακριβώσουμε και με αριθμητικά στοιχεία. Γιατί έτσι γίνεται καλύτερα αντιληπτή κατάσταση. Ότι οι επενδύσεις που έρχονται από την Ευρώπη στη Λατινική Αμερική είναι επενδύσεις που έρχονται για να μείνουν. Είναι greenfield όπως λέμε. Είναι επενδύσεις που δεν αποκτά μόνο ε, ε, περιουσιακά στοιχεία, αλλά δημιουργεί και παραγωγικότητα. Το 60% των εξεγγελθέντων σχεδίων της και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, Λατινική Αμερική είναι κυρίως στη Βραζιλία και έχουν και ένα σκέλος ε, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που ενισχύουν τη μεταφορά τεχνολογίας και ως εκ τούτου αξιοποιούν καλύτερα το δυναμικό, το ανθρώπινο δυναμικό, ε, συμβάλλουν στην αύξηση των μισθών και στην ε, καινοτομία και παραγωγικότητα. Και οι περισσότερες ευρωπαϊκές επενδύσεις στόχο έχουν τη δημιουργία νέων παραγωγικών δυνατοτήτων με ένταση γνώσης και ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι αυτή η νέα ε, παραγωγική αυτό το νέο παραγωγικό δυναμικό θα πρέπει να το ενισχύσουμε και χάρη στη συνεργασία και τη βοήθεια των βουλευτών, στη βοήθεια, χάρη στη βοήθεια της κοινωνίας των πολιτών, θα έχουμε ένα σημαντικό αντίκτυπο. Στην Λατινική Αμερική έχουμε δύο βασικά εργοστάσια ανισοτήτων. Το ένα ε, οφείλεται στην αδυναμία απορρόφησης της τεχνολογικής ανάπτυξης. Δεν είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα ικανότητας αντίληψης αλλά και απορρόφησης της τεχνολογικής πρόοδου. Δεύτερο εργοστάσιο ανισοτήτων είναι η παραγωγική ετερογένεια. Έχουμε διάφορες επιχειρήσεις μεγάλης, μεσαίας και μικρής παραγωγικότητας, αλλά δυστυχώς οι περισσότερες είναι επιχειρήσεις χαμηλής παραγωγικότητας. Ο Επίτροπο Σταγιάννη μίλησε για το δυναμικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και στη Λατινική Αμερική οι μικρομεσαίε επιχειρήσει παράγουν το 60% των θέσεων απασχόληση. Αλλά οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, το 70% των μικροεπιχειρήσεων, δεν έχουν καν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό πραγματικά είναι τραγικό για τη σήμερα ημέρα και το 70% το 7% των, των επιχειρήσεων της Λατινικής Αμερικής ε, πραγματοποιούν ηλεκτρονικά τι εργασίες του. Ε, υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα και ψηφιακό. Δεν είναι μόνο να φτάσει η τεχνολογία σε εμά, αλλά να μπορέσουμε και να την απορροφήσουμε αυτή τη τεχνολογική πρόοδο. Και αυτή η γεφύρωση των κενών και του χάσματος μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι σημαντική, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η κινητήρη μοχλή της ανταγωνιστικότητας. Θα πρέπει λοιπόν να απορροφήσουμε καλύτερα τη τεχνολογία για να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσει να βελτιώσουν το δυναμικό του και να έχουν καλύτερη πρόσβαση και στην πίστη, στο δάνειο. Ε, η Χιλή διοργανώνει με μεγάλη φροντίδα την επόμενη σύνοδο κορυφή και έχουμε μαζί μα και εκπροσώπους τη Χιλή και τον βουλευτή Πισάρο και προσπαθούμε όλοι να βοηθήσουμε τη Χιλή για να σταθεί με επιτυχία αυτή η σύνοδο κορυφή και να μεταφέρει διαφορετικά μηνύματα αυτή τη φορά. Μηνύματα που θα ε, δείχνουν ότι κοινό μας κεκτημένο είναι να πραγματοποιήσουμε το όνειρό μας για μία ε, ανάπτυξη αηφόρο αλλά με ισότητα, με ισότιμα δικαιώματα, ε, με επαναπροσδιορισμό των αξιών μας και των διαφόρων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής και με την Ευρώπη σημαντικό μας εταίρο για την πραγματοποίηση του ονείρου μας. Και σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές βλέπουμε με διάβια ότι κάθε περιοχή έχει τις δικές της προκλήσεις και τις δικές της ευθύνες. Από τη μια όχθη του Ατλαντικού ε, πρόκληση είναι να διασφαλιστεί η ευημερία, να διατηρηθεί και να μην χαθεί. Και από την άλλη όχθη η κατάκτηση αυτής της ευημερία και η διεύρυνσή της ώστε να είναι προσιτή σε όλους. Είναι διαφορετικές λοιπόν οι προκλήσεις μας. Αλλά εμείς προσβλέπουμε ε, και η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική όπως και η Ευρώπη να γίνουν οι περιοχές του κόσμου όπου θα συνδυάζεται η δημοκρατία με την ελευθερία, με την ευημερία και την κοινωνική ένταξη. Γιατί θέλουμε να γεφυρώσουμε τα κενά και τα χάσματα. Θέλουμε να γεφυρώσουμε αυτά τα χάσματα στη Λατινική Αμερική και θέλουμε σε αυτό το στόχο προνομιακός μας εταίρος να είναι η Ευρώπη, γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι και στη Λατινική Αμερική έφτασε η ώρα της ισότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Αλήθεια Μπάρσενα. Πραγματικά πολύ εμπνευσμένη η ομιλία σου. Το λόγο έχει τώρα η συμπρόεδρος της συνέλευσης, η κυρία Γκλώρια Ορκελή. Μετά από τόσες πληροφορίες και τόσο σημαντικά στοιχεία και τόσο εντυπωσιακές ομιλίες, θα καταβάλω κι εγώ ε, μία προσπάθεια, γιατί από εδώ έχω και καλή θέα και βλέπω ποιος κοιμάται. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω τον ενθουσιώδη χαιρετισμό της α, λατινικής συνιστώσης της, της συνέλευσης και να μεταφέρω έναν θερμό χαιρετισμό εκ μέρους της α, όμορφης και αξιοπρεπούς Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής προς την Ευρώπη. Είναι αναφυσβήτητο ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Έχουμε μια αλλαγή εποχής πραγματικά. Ε, και στην Λατινική Αμερική και στην Ευρώπη αντιμετωπίζουμε υπερβατικές πραγματικότητες και σημαντικές προκλήσεις. Η Λατινική Αμερική, η Λατινική Αμερική δεν είναι πια μια ιστορική έννοια. Έχει μετατραπεί σε μια πολιτική και οικονομική πραγματικότητα που έχει σημαντική επιρροή και συνέπειες και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη παγκοσμίω. Και σε λίγες μέρες θα συστηθεί στο Καράκα της Βενεζουέλας η κοινότητα των ε, Λατινοαμερικανικών και χωρών της Καραϊβικής, η ΣΕΛΑΚ, μια απόφαση που ελήφθη το 2010 στη Σύνοδο Κορυφής του Κανκού στο Μεξικό. Χωρίς παρέμβαση α, ε, δυνάμεων και υπεροπτικών τάσεων θα αναζητήσουμε και θα προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε το κοινό μας μέλλον. Και είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτή η περιοχή μας, όχι ως ομάδα αντικρώμενων συμφερόντων, αλλά ως το απάβγασμα της του ιστορικού πλούτου των λαών μας και της οριμότητας που επιτύχαμε προκειμένου να υλοποιήσουμε τα κοινά μας συμφέροντα. Η ΣΕΛΑΚ θα γίνει ένα κοινό εργαλείο για να ικανοποιήσουμε τα κοινά μας συμφέροντα και ενδιαφέροντα και πιστεύω ότι μπορεί μερικοί επικριτές ε, ή αντίπαλοι μας να κρίνουν όσο τοπικά τα σχόλιά μου, αλλά νομίζω ότι η δέσμευσή μας είναι για περισσότερη ισχύ, και ενότητα. Πολλοί ητοπαθείς και μυρολάτρες ε, φορείς του ιού της απόσχησης και της ενότητας βλέπουν την ενότητα της Λατινικής Αμερικής ως ψευδέστηση, ως οφθαλμαπάτη, ως ουτοπία, ως φάτα μορκάνα και αυτοί που είναι κατά της ενότητας και σπέρνουν ζυζάνια θα κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφύγουν αυτή την πραγμάτωση της ενότητας στη Λατινική Αμερική. Γι' αυτό θα ήθελα να επιμείνω ότι βρισκόμαστε σε, μια, σε ένα μετέχμιο, σε μια αλλαγή εποχής όπου οι προοδευτικές κυβερνήσεις ε, αναλαμβάνουν τα ενία της εξουσίας με σημαντική λαϊκή υποστήριξη και κυρίως επιδεικνύοντας αλληλεγγύη. Όπως είπε η Γιωκόντα Βέλη, η Νικαραγωνή συγγραφέας, η αλληλεγγύη είναι η τρυφερότητα των λαών. Κατά τη γνώμη μας, ε, οι σχέσεις μεταξύ των χωρών θα πρέπει να έχουν ως θεμέλια το σεβασμό, την αξιοπρέπεια, την αυτοδιάθεση και την κυριαρχία. Αναφυσβήτητα, οι διάφοροι πόλεμοι, οι σημερινοί πόλεμοι και οι οι διάφορες εισβολές που εκπορεύονται από την απληστία, από τον νεοπικρατικό χαρακτήρα, από τον καταναλωτισμό είναι σενάρια που με την συνενοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης φτάνουν στα, στις αιστείες μας ως τετελεσμένα γεγονότα και αυτά μπροστά στην ε, γενική αδιαφορία. Αυτό δημιουργεί μια επικίνδυνη κατάσταση όπου οι ίδιοι λαοί μας μπορούν να είναι τα επόμενα θύματα του αυταρχισμού και της αυθαιρεσίας. Ταυτόχρονα όμως μια τέτοια κατάσταση κρούει τον κόδωνα του κινδύνου Δημιουργείται μια παγκοσμιοποίηση της διαμαρτυρίας με δραστήριο αλλά ειρηνικό τρόπο. Είχαμε την, την Αραβική Άνοιξη, το κίνημα των αγανακτισμένων και το κίνημα είμαστε το 99%. Η νομιμοποίηση και η αντιπροσωπευτικότητα των εκλεγμένων βουλευτών μας ε, δημιουργεί τη δέσμευση της αναχέτησης όλων των ανταρτικών και αποσχιστικών τάσεων στον κόσμο. Και Επίσης μας δίνει την ευκαιρία για μια ενυφάλια, ορθολογική και ρεαλιστική ανάλυση των οικονομικών και κοινωνικών συστημάτων και των δημιουργικών και ευρηματικών εναλλακτικών λύσεων. Στη Eurolat, βασικός μας στόχος είναι να ενισχύσουμε την δημοκρατική εκπροσώπηση των λατινοαμερικανικών και ευρωπαϊκών λαών στην διαδικασία της διπεριφερειακής στρατηγικής σύνδεσης και συνεργασίας. Ο πλούτος μας έγκυται στην πολυμορφία μας. Έχουμε ανοιχτές συζητήσεις, πλουραλιστικές, συμμετοχικές και πραγματικά ειλικρινείς. Γι' αυτό και η Eurolat είναι μια εξόχως δημοκρατική κοινοβουλευτική συνέλευση που θα αποτελέσει το φυτόριο ευρηματικών προτάσεων και αποφασιστικότητας και θα συμβάλλει ώστε διάφορα θέματα διπεριφερειακής συνεργασίας ε, θα καταλήξουν σε αποφάσεις που θα ωφελήσουν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού που εκπροσωπούμε. Και έτσι θα μπορέσουμε να κληροδοτήσουμε στις επερχόμενες γενναίες έναν καλύτερο κόσμο. Έχουμε πραγματικά στην Κυρολάτη ένα ιδεώδες εργαλείο για να προωθήσουμε τις ε, συναλλαγές μας και να έχουμε διάλογο με βάση την αρχή της ισότητας και της ισοτιμίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής και προκειμένου να ε, κατακτήσουμε αυτή την ισότητα και την ισοτιμία και στις περιφέρειες και στις ε, χώρες και στις κοινωνίες μας δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τις ασυμμετρίες και τις ανισότητες που χαρακτήρισαν τον ιστορικό συσχετισμό και τη διασύνδεση των δύο υπήρων. Τώρα ο μόνος τρόπος για να υλοποιήσουμε ε, επιτυχείς προσπάθειες είναι να έχουμε αξιοπρεπή και δημοκρατική διπεριφερειακή ολοκλήρωση με σεβασμό, διάλογο, ανοχή και συνενετική συνεργασία. Τα πρώτα αυτά χρόνια περάσαμε από τη φάση των θεμελίων στην πλήρη αντίληψη των αρχών που θα μας επιτρέψουν να αναγνωρίσουμε και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες, να άρουμε τα εμπόδια και να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Για να προχωρήσουμε σε αυτή τη μοναδική ευκαιρία δημοκρατι... κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που προβλέπει συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων και δίνει, δίνει, είναι υπόλογη απέναντι στους πολίτες, επιτρέπει τη λογοδοσία και την υπευθυνότητα απέναντι στις κοινωνίες μας. Είμαστε βαθύτατα πεπισμένοι ότι ο σεβασμός των σχέσεών μας και ο σεβασμός των δικαιωμάτων μας θα συμβάλλουν αναφίβολα στην ειρήνη και στην ευημερία. Παρα, παραφράζοντας ε, τον ε, κορυφαίο Μπενίτο Σουάρες πριν από 140 χρόνια μεταξύ εθνών και ανθρώπων το ο σεβασμός του δικαιώματος του άλλου είναι αυτό που δημιουργεί την ειρήνη. Ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της Ευρώ ε, Λατινοαμερικανικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Σας ευχαριστούμε, Γκλώρια Ορκελή. Η αλήθεια είναι ότι ήταν τόσο εμπνευσμένε και καταπληκτικές οι ομιλίες των προλαλισάντων, κάτι που με διευκολύνει και εμένα. Και θα ήθελα να πω ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και σε ένα κλειδί του δικού μας χρονο... σε ένα σημείο κλειδί του δικού μας χρονοδιαγράμματος. Ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διανύει μια οικονομική, πολιτική, κοινωνική κρίση, αλλά και μια κρίση εμπιστοσύνη. Και ε, υπό, αυτό το πρίσμα και με μεγάλη μετριοφροσύνη θα ήθελα να σας ε, επισημάνω ένα από τα θέματα που ήταν ένα από τα κορυφαία θέματα της ε, διάσκεψης κορυφής της Ασουνθιών. Αφορούσε τα αναπτυξιακά μοντέλα και τη τις μεταρρυθμίσεις ε, στις διάφορες χώρες. Ο Αντιπρόεδρος τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Σταγιάννη, μα είπε το πρωί ότι δεν έχει πεθάνει, ούτε έχει ταφεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το αναπτυξιακό μοντέλο που εφαρμόσαμε μας ε, έφερε στο επίκεντρο τις αξίε. Είναι ένα σχέδιο που στηρίζεται στην ειρήνη, την ε, κατανόηση, την ομόνοια, την αλληλεγγύη και ταυτόχρονα είναι ένα μοντέλο με απτές πρόοδους με αυτά επιτεύγματα και κατορθώματα που μετατράπηκαν σε προδιαγραφές κοινωνικής πρόοδου άνευ προηγουμένως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα παράγουμε το 1 τρίτο του παγκόσμιου ΑΕΠ. Έχουμε εδραιώσει μια ενιαία αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών με 300 εκατομμύρια που χρησιμοποιούν το κοινό νόμισμα Είμαστε πρώτο εισαγωγέ και εξαγωγέ αγαθών και υπηρεσιών, βασικό παγκοσμίω δωρητή αναπτυξιακή βοήθεια ε, και στοχο μα είναι να γίνουμε και σημαντικό πολιτικό εταίρο στην παγκόσμια σκηνή. Μιλήσαμε πολλά, ε, πολύ για το BRICS και στην, Ευρωπαϊκή, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα συζητηθεί μία έκθεση ενός βουλευτή της πολιτικής μου ομάδας για τις χώρες BRICS με συγκεκριμένη κατεύθυνση πολύ οξυδερκή αντιμετώπιση. Θα ήθελα να σχολιάσω και εγώ κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά την παρουσία μερικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγοι γνωρίζουν ότι η Αυστρία, για παράδειγμα, η πατρίδα της ε, Μπένιτα Φερέρο, ε, ε, υποδέχεται διπλάσιο ρυθμό μεταναστών από τη Βραζιλία. Η, η Δανία που έχει εμπόριο υπηρεσιών μεγαλύτερο από τη Ρωσία. Η Σλοβενία έχει τριπλάσιες αθλητικές επιτυχίες από την Ινδία. Ή το Λουξεμβούργο, 350.000 ε, πολίτες, έχει περισσότερα στρατεύματα από την Κίνα σε παγκόσμιες ενέργειες. Και η Ελλάδα έχει τριπλάσια επιστημονική συμμετοχή από την Νότια Αφρική σε παγκόσμιε οργανώσει, παρά τη δινή οικονομική τη κατάσταση. Βλέπετε ότι ακόμη και μικρέ χώρε ε, συμβάλλουν ε, και έχουν σημαντική παρουσία σε διάφορου τομεί. Και πιστεύω ότι με ενίσχυση τη συνεργασία μα ε, η παρουσία αυτή θα γίνει ακόμη πιο αισθητή. Βέβαια, αυτό είναι ένα στιγμιότυπο Υπάρχουν όμως κάποιες τάσεις και σίγουρα υπάρχει μια μετατόπιση του παγκόσμιου οικονομικού άξονα από τον Ατλαντικό προς τον Ειρηνικό και Ινδικό ωκεανό. Εμείς φυσικά έχουμε και το οικονομικό και νομισματικό μας σχέδιο που είχε κάποιες αδυναμίες στην στο σχεδιασμό του και έχουμε και ένα τεράστιο έλλειμμα στην οικονομική διακυβέρνηση υφιστάμε αυτή τη στιγμή τις αδυναμίες αυτού του σχεδίου. Εμείς παρόλα αυτά είμαστε πολίτες μιας ένωσης και εδώ έχουμε ένα ποιοτικό άλμα από την ε, Ένωση των Καταναλωτών στην Ένωση των Πολιτών. Μια Ένωση των Πολιτών όμως προϋποθέτει ε, ένα κοινοβούλιο που καλείται να κυρώσει όλες αυτές τις συμφωνίες που μας ανέφερε ο Αντιπρόεδρος Κολομβίας, ο κύριος Γαρθών. Ένα άλλο σημαντικό θέμα ανέφερε η Αλίσσα Μπάρσενα στην πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία της είναι το θέμα των υποδομών γιατί η ολοκλήρωση δεν είναι μόνο νομική και πολιτική έννοια. Είναι εξόχως υλική, πραγματική. Και οι υποδομές, παρόλο που είναι ε, μόνιμα πάγιες δομές, πολλές φορές συμβάλλουν στις καθυστερήσεις. Άλλο σημαντικός φορέας πρόοδου είναι η παιδεία ή ε, το θέμα των πρώτων υλών. Η, πρώτη η σημαντικότερη πρώτη ύλη είναι η θεά ύλη, είναι η θεά ουσία του κεφάλου, γιατί το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό που συμβάλλει στην έρευνα και στην τεχνολογική ανάπτυξη. Πριν από 40 χώρες, πριν από 40 χρόνια, συγγνώμη, χώρες όπως το Μεξικό, η Βραζιλία ή η Βενεζουέλα είχαν εισόδημα δεκαπλάσιο από την Νότια Κορέα. Σήμερα έχει αντιστραφεί αυτή η βενεζουελα ειχαν εισοδημα δεκαπλασιο απο τη νοτια κορεα σημερα εχει αντιστραφει αυτη η ταση και η Νότια Κορέα έχει διπλάσιο εισόδημα από τη Βενεζουέλα ή το Μεξικό για παράδειγμα. Είναι απίστευτο το, στοιχείο, το, το στοιχείο για την ανανέωση των διπλωμάτων ευρυστεχνίας. Ε, ετησίως η Νότια Κορέα καταθέτει 800.000 διπλω, ε, διπλωμάτων ευρυστεχνίας από τις, από, τις, από τις λατινοαμερικανικές χώρες η Βραζιλία έχει τις μεγαλύτερες επιδόσεις με 100 μόνο αιτήσει διπλωμάτων ευρυσιτεχνίας το χρόνο το Μεξικό 53 και η Αργεντινή 30 αιτήσει. βλέπετε τεράστια διαφορά μεταξύ των διπλωμάτων ευρυσιτεχνίας μεταξύ Ασίας και Λατινικής Αμερικής μετά από 60 περίπου χρόνια διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκληρώσης αυτό που μπορούμε να σας πούμε στην Ευρώπη είναι ότι η αηφόρος ανάπτυξη ε, δεν θα είναι εύκολη χωρίς ολοκλήρωση. Αυτή είναι η δική μας εμπειρία. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοούμε ή αδιαφορούμε για τις δυσκολίες ή ότι θελοτεφλούμε, γιατί σήμερα ακριβώς βιώνουμε αυτές τις δυσκολίες της διαδικασίας ολοκλήρωσης. Γνωρίζουμε όμως ότι η επιτυχία του μοντέλου μας στηρίχθηκε στην ολοκλήρωση. Και μάλιστα η ολοκλήρωση είναι πολύ πιο σημαντική στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Δεν πρόκειται να σας κουράσω άλλο. Θα ήθελα απλώς να σας πω ότι όταν περάσει αυτή η περίοδος και όταν ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική θητεία του 2014 θα εορτάζουμε ένα αιώνα μετά το Μεγάλο Πόλεμο που τον ακολούθησε ένας άλλος ζωφερός πόλεμος, μία από τις πιο σκοτεινές ιστορίες της Ευρωπαϊ... Ε, σελίδες της ευρωπαϊκής ιστορίας. Και το σημερικό σενάριο ήταν πραγματικά διανόητο πριν από μερικά χρόνια. Είμαστε πολύ περήφανοι και για τον πολιτισμό μας και ε, για την κουλτούρα μας, για τις κοινέ αξίες που έχουμε με τη Λατινική Αμερική και θα ήθελα να σας πω ότι η ευρωπαϊκή ιστορία είναι μια ιστορία υπέρβασης των δυσκολιών. Αναφέρθηκε ότι η Ευρώπη ε, κινητοποιείται με την αναγκαιότητα και μόνο όταν αναγκαιότητα φτάνει προ, προ πυλών καταφέρνει και κάνει ένα ποιοτικό άλμα. Είχαμε πριν από μερικά χρόνια τη, το 70 τον ευρωσκεπτικισμό, τη δεκαετία του 80 είχαμε την ενιαία αγορά και το νέο όριο ήταν η Ευρώπη χωρίς σύνορα και σας διαβεβαιώ ότι δεν θα εγκαταλείψουμε αυτό το σχέδιο. Αυτό το σχέδιο που έχει αρχίσει και εκρήγνεται στις διάφορες ραφές. Δεν θα το εγκαταλείψουμε, θα προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και ευελπιστώ ότι στις ημερίδες που θα έχουμε με τις διάφορες επιτροπές θα λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην παγκόσμια σκηνή. Η Αλήσια Μπάρσενας μίλησε για την εμφάνιση της Κίνας. Τα στοιχεία πραγματικά είναι απίστευτα. Με βάση το Κινέζικο ε, Υπουργείο Εμπορίου το πρώτο τρίμηνο του 2011 αυξήθηκαν οι κινέζικες εξαγωγές προς τη Λατινική Αμερική κατά 40 και τα 100, 49 δις περίπου ε, δολάρια, κάτι που δείχνει την ανάγκη ισορροπημένων παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών που δεν θα ε, περιορίζονται μόνο στις πρώτες ύλες, αλλά θα καλύπτουν και τα μεταποιημένα προϊόντα. Σας ευχαριστώ. Καλή εργασία σας, εύχομαι και καλή συνέχεια. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και σε 11.30 η Μαρία Μεχία θα κάνει μια δήλωση και θα ακολουθήσει συζήτηση με τα μέλη της συνέλευσης. Ευχαριστώ. Περνάμε στην επόμενη φάση των εργασιών μας. Τους Θέρμα παρακαλώ τα μέλη να καθίσουν, να λάβουν θέσεις. Θα είμαστε πολύ αυστηροί στη χορήγηση του χρόνου αγόρευσης, γι' αυτό και ζητώ την κατανόησή σας εκ των προτέρων. Να σας εξηγήσω καταρχήν τη μεθοδολογία. Θα ακούσουμε τη δήλωση και μετά θα έχουμε γύρους τριών ομιλητών για να μπορούμε να ακούμε και τις απαντήσεις. Ευτυχώς ρολόι έχουμε, θα τηρούμε το χρόνο αυστηρά και μετά προς το τέλος συνεδρίασης θα βγάλουμε και την ιστορική οικογενειακή φωτογραφία. Η Γενική Γραμματέας της Σούρ είναι μια νέα πανέξυπνη και πανέμορφη γυναίκα. Ξέρω ότι ω άνδρα ήταν κάπω δύσκολο να κάνει τέτοια σχόλια κανεί. Εγώ ω γυναίκα, εκπροσωπώντα και την γυναικεία, και την ανδρική οπτική, μπορώ να κάνω αυτέ τι φιλοφρονήσει προ την ε, Γενική Γραμματέα τη Ένωση Νοτιοαμερικανικών Εθνών, τη UNOSUR, την κυρία Μαρία Έμα Μεχία Βέλεφ. Η κυρία Μεχία ανέλαβε τη Γενική Γραμματεία της UNASUR στις 11 Μαρτίου του 2011. Προηγουμένως ε, τελε, διατέλεσε Υπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας μεταξύ Ιουλίου του 1996 και Μαρτίου του 1998 επί Σαμπέρ Πισάρ, Προέδρου της Κολομβίας. Θα γνωρίζετε, ήταν δύσκολη εκείνη η εποχή για την Κολομβία και σήμερα ακούσαμε τη σημαντική πρόοδο επιτέλεση στο μεταξύ αυτή η χώρα. Η κυρία Μεχία θα μας μιλήσει σήμερα όχι μόνο εκ μέρου της πατρίδας της, της Κολομβίας, αλλά θα μας μιλήσει και για τις 12 χώρες της Γιουνοσούρ που εκπροσωπούν το 70% του πληθυσμού της Λατινικής Αμερικής, 400 εκατομμύρια κατοίκους περίπου. Αυτή τη στιγμή και με την τεράστια αυτή πολυμορφία της Λατινικής Αμερικής προσπαθούμε να διαμορφώσουμε μια κοινή ταυτότητα και κοινή λατινοαμερικανική ηθαγένεια. Και γι' αυτό ε, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε και ένα χώρο χωρίς σύνορα για να επιτρέψουμε καλύτερα την ολοκλήρωση. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα από κανέναν ότι όταν καταργούνται τα σύνορα αναφαίνονται διάφορα άλλα προβλήματα και αυτό θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε σήμερα με την ε, έκθεση αυτή. Πάντως ε, έχουμε παρατηρήσει αύξηση της κατανάλωσης κοκαίνης και λεύκασης χρήματος μεταξύ άλλων. Αυτά τα προβλήματα εξετάζει η UNASUR και έχουμε και το πρώτο πρόγραμμα, αεροναυπηγικό πρόγραμμα της Λατινικής Αμερικής και εξετάζουμε και τα στάδια υλοποίησης των διαφόρων προγραμμάτων υποδομή και ενεργειακών προγραμμάτων και σχεδίων. Χωρί άλλη χρονοτριβή, θα δώσω το λόγο στην Μαρία Έμα Μεχία Βέλεθ και την καλωσορίζω επί τη ευκαιρία. Σα ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για την φιλοξενία σας αυτή και για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω την Ένωση Λατινοαμερικανικών Εθνών, τη UNASUR, Ευχαριστώ και την Πενίτα για την παρέμβαση που έκανε προηγουμένως. Εσείς θα βρεθείτε στην πρώτη γραμμή αυτών των προσπαθειών, χάρη στο Ίδρυμά σας και θα δρέψουμε τους καρπούς αυτής της συμμαχίας. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο και όπως ακούσαμε και το πρωί έχουμε πολύ σημαντικές ευκαιρίες συνάντησης σε μια πραγματικά δύσκολη συγκυρία για την ε, ζωή και την καθημερινότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσφατα η Άγγελα Μέρχελ χαρακτήρισε την εποχή αυτή τη πιο δύσκολη εποχή ίσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αυτό το μήνυμα πραγματικά μας εντυπωσίασε όλους. Ήμουνα πρόσφατα στη Μαδρίτη για την τρίτη διάσκεψη παγκόσμιας πρόοδου και είπαμε ότι ο κόσμος ε, δεν έχει την πολυτέλεια να επιτρέψει ε, να, να βαγίσει το ευρωπαϊκό σχέδιο γιατί αποτελεί πια η Ευρωπαϊκή Ένωση τμήμα της δημοκρατικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και ε, συμβολίζει τις κοινέ μας αξίες όπως μας είπε ο κύριος Αλαφράγκα. Η Λατινική Αμερική ε, ζει πολύ θετική συγκυρία και εδώ και τρεις, μήνες και, τρία χρόνια και έξι μήνες για πρώτη φορά ε, υπογράφηκε η συντακτική συνθήκη της Γιουνασούρ μια νέα φάση ολοκλήρωσης και από τη Βραζίλια το 2008 μέχρι σήμερα διανύσαμε πολύ σημαντική πρόοδο και παρά τις ιδεολογικές μας διαφορές ή διαφορές ε, αναπτυξιακού μοντέλου που εφαρμόζουμε οι οικονομικές διαφορές καταφέραμε παρόλα αυτά να καταλήξουμε σε πολύ σημαντικές συμφωνίες στη Λατινική Αμερική. Όταν δέχτηκα την πρόσκλησή σας, κύριε Ιγνάσιο Σαλαφράγκα και κυρία Γκλώρια Οκελή, σκέφτηκα ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η ευκαιρία και πραγματικά γίνεται ένα κλικ με αυτή την κατάσταση, γιατί για πρώτη φορά αρχίζουμε και σκεφτόμαστε για το κοινό μας πεπρωμένο και μάλιστα σε μία ήπειρο που ασχολήθηκε τόσο πολύ με τη διαδικασία ολοκλήρωσης εδώ και 200 χρόνια ε, θα γιορτάσουμε μάλιστα και τους δύο αιώνες αυτής της προσπάθειας διαπιστώνουμε μετά ε, τις δυσκολίες ε, του 19ου αιώνα και μετά τον κύκλο του, των πολέμων του 20ου αιώνα μετά είχαμε τη συνένεση της Ουάσιγκτον, το τέλος του ψυχρού πολέμου, όπως μας είπε και η πρόεδρος Οκελή. Και αυτή η ιδέα, αυτό το σχέδιο της ολοκλήρωσης ε, ποτέ δεν αποδυναμώθηκε, ποτέ δεν εξανεμίστηκε. Απλώς στράφηκε περισσότερο προς το εμπορικό σκέλος αφήνοντας κατά μέρους το πολιτικό. Και εσείς καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο γνωρίζετε γιατί το βιώσατε ε, η ΑΛΑΚΑ έγινε ΑΛΑΝΤΙ, Ευρωπαϊκή Κοινότητα των Άνδεων, περάσαμε στη Μερκοσούρ, πολύ σημαντικές διαπεριφερειακές προσπάθειες και στόχος μας είναι η όλο και μεγαλύτερη ολοκλήρωση στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική. Πάντως από το 2000 όταν ο Φερνάντο Ερίκε Καρδόσο συγκάλεσε για πρώτη φορά τους προέδρους ε, της Λατινικής Αμερικής ε, σε κοινή συνεδρίαση, ξεκίνησε η συζήτηση για την ολοκλήρωση. Μία συζήτηση που ξεκίνησε υπό χαλεπές πολιτικές συνθήκες, γιατί ξεκίνησε η συζήτηση λίγο μετά την ε, εισβολή των κολοβιανών στρατευμάτων στην, στον Ισημερινό μετά, για να κλείσουν το καταβλισμό της ΦΑΡΚ. Μετά είχαμε την, το σύμφωνο της Αντακρούς στη Βολιβία και το δημοψήφισμα για το αυτόνομο καθεστώς, κάτι που δημιούργησε μεγάλες τάσεις. Και μάλιστα η Μπατσελέτ ε, κάλεσε κοινή συνεδρίαση για να αποφευθεί η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή και υπήρχαν και διάφορες άλλες ε, εντάσεις και τριβές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και της περιοχής εξαιτίας της ε, στρατιωτικής παρουσίας των Αμερικανών στις ε, βάσεις της Κολομβίας. Με όλη αυτή την αντίξωη κατάσταση ήταν ζωφερές οι προβλέψεις για το μέλλον του Μερκοσούρ. Παρ' όλα αυτά, χάρη στον πολιτικό διάλογο, και χάρη στον προκατοχό μου Ερνέστο Κίσνερ, τον ε, πρώην πρόεδρο, δώσαμε έμφαση σε αυτή την ολοκλήρωση και πριν από 15 μήνες περίπου ε, ευτυχώς εξομαλήθηκε η κατάσταση μεταξύ Βενεζουέλας και Κολομβίας και σήμερα υπάρχει μια υγιής κατάσταση, μια πολύ ομαλή και ήρεμη και διαμορφώνεται πια η Λατινική Αμερική ως ζώνη ειρήνης, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Όπως ε, είχαμε και το Νοτιοαμερικανικό Συμβούλιο Άμυνας, μια άλλη πρωτοβουλία που ε, εμπεδώνεται όλο και περισσότερο και στην τελευταία συνεδρίαση που είχε το Συμβούλιο αυτό πριν από 10 μέρες στη Λίμα, εγκρίναμε μια κοινή μεθοδολογία για το μετριασμό των στρατιωτικών δαπανών και το στρατιωτικό δυναμικό των χωρών μελών και το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει κάποια μέτρα με βέση εμπιστοσύνη. Και μάλιστα η Γερμανία μα υποστήριξε πολύ σε αυτό το πολύ σημαντικό έργο άμυνα. Δημιουργήθηκε και το Κέντρο Στρατηγικών Αμυντικών Σπουδών για να επεξεργαστεί κάποια ε, δόγματα και θεωρίες σε συνεργασία με ε, στρατιωτικούς αλλά και με τα αρμόδια υπουργεία. Το κέντρο αυτό βρίσκεται στο Buenos Aires. Έχουμε λοιπόν μια ζώνη ειρήνης σε μια ε, περιοχή που είναι η μόνη αποπυρηνικοποιημένη περιοχή. Μόνο το 32 ήταν ο τελευταίος μας πόλεμος ε, στη Βολιβία, γιατί μιλούμε για τις επαιτίους και τις δύσκολες περιόδους αυτές, τη δύσκολη αυτή περίοδο για την Ευρώπη. Εμείς ήμασταν πραγματικά ε, μια περιοχή ελεύθερη από πολέμους. Είχαμε μόνο κάποιες διμερείς τριβές μεταξύ όμορων χωρών, αλλά όχι πραγματικούς πολέμους. Στη Λατινική Αμερική έχει, δημιουργείται ένα θεμελιώδες πρόβλημα τώρα τελευταία με τους φυσικούς πόρους. Το είπε και η Αλίσια το πρωί. Η Αλήσια μας είπε το πρωί ότι έχουμε πέντε από τις χώρες με τη μεγαλύτερη βιοπικιλιομορφία, έχουμε το 1 τρίτο του παγκόσμιου, του παγκόσμιου αποθέματος ύδατος, έχουμε 30% ε, των δασών, έχουμε τεράστια κοιτάσματα και ορυκτού πλούτου και φυσικά επισητιστικά αποθέματα. Για το 2025 θα έλεγα ότι το 40% των τροφίμων παγκοσμίω θα προέρχονται από τη Λατινική Αμερική. Διανύουμε παρόλα αυτά μια δύσκολη κατάσταση και ε, ευτυχώς ξεπεράσαμε την κρίση του 2008. Τη βιώνουμε βέβαια αλλά πολύ πιο ήπια πια. Και την Παρασκευή στις 25 του μηνός θα έχουμε στον Πόνο Σάιρες το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών και Κεντρικών Τραπεζών της Λατινική Αμερική. Και ελπίζουμε ότι θα προσανατολιστούμε σε τρεις βασικούς άξονες. Καταρχήν, διαφύλαξη των νομισματικών μας αποθεμάτων μεταξύ 600 και 700 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθόλου αμεληταίο ποσό για νομισματικό απόθεμα, γιατί όπως λένε και οι πρόεδροι μας, ε, αξίζουμε πραγματικά να διεκδικήσουμε μεγαλύτερη παρουσία και, και αντιπροσωπευτικότητα στο παγκόσμιο νομισματικό σύστημα. Ε, το ακούσαμε πρόσφατα και στις Κάνες. Επίσης θέλουμε να ενισχύσουμε το Λατινοαμερικανικό Ταμείο Αποθεμάτων και ε, ενίσχυση της Λατινοαμερικανικής ε, Τράπεζας Ανάπτυξης και της Τράπεζας των Άνδεων. Εκεί οι βασικοί διοικητές, οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών θα συζητήσουμε τους Υπουργούς Οικονομικών όλα αυτά τα θέματα και θα βελτιώσουμε τις ανταλλαγές μεταξύ και τοπικών νομισμάτων. Είχαμε το παράδειγμα της Βραζιλίας και της Αργεντινής. Αυτό το παράδειγμα μπορούμε να το μιμηθούμε και σε άλλες περιοχές της Λατινικής Αμερικής και θέλουμε φυσικά να διευρύνουμε και το διαπεριφερειακό εμπόριο που αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο 25%. Για μας ε, δεν ήταν καθόλου εύκολο αυτό το διαπεριφερειακό εμπόριο γιατί είναι πολύ πιο εύκολο ε, να εξάγουμε εκτός ε, Λατινικής Αμερικής να περάσουμε τον ωκεανό παρά να περνάμε τις οροσυρές των Άνδεων και να έχουμε εξαγωγές σε γειτονικέ χώρες. Το πρωί ακούσαμε πως μεταξύ του 80 και του 2003 ε, είχαμε 38 οικονομικές κρίσεις στη Λατινική Αμερική και μάλιστα αντλήσαμε πολλά διδάγματα από τα παθήματα αυτά και όπως είπαμε στο G20 έχουμε και την BRICS στην οποία συμμετέχει η Βραζιλία και το σύμπλη που θα είναι το BRICS του 21ου αιώνα. Και η Κολομβία συμμετέχει σε αυτή τη δεύτερη ομάδα. Τα τελευταία 15 χρόνια περάσαμε από το 6% στο 24% του εμπορίου νότου-νότου. Βέβαια, ακούσαμε για τη σημαντική και ανερχόμενη παρουσία της Κίνας και όπως είπατε και εσείς, αυτό το πρώτο τρίμηνο του 2011 το εμπόριο αυξήθηκε κατά 44%. Δηλαδή, 40 ε, δισεκατομμύρια ευρώ και μάλιστα αναφέρθηκε ε, στη ΣΕΠΑΛ ότι η Κίνα πριν το 2015 θα μετατραπεί στο δεύτερο σημαντικό εταίρο μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, η ανάπτυξη κυμαίνεται μεταξύ στο 4 και το 5% για τα επόμενα χρόνια στη Λατινική Αμερική. Βέβαια υπάρχει μεγάλη διαφορά στις σχέσεις μεταξύ Λατινικής Αμερικής και Κίνας και Λατινικής Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει διαφορά και ως προς το διαπεριφερειακό εμπόριο. Αναφέρθηκε σημαντικό, ναι, αναφέρθηκε το σημαντικό θέμα των υποδομών σε ό,τι αφορά τη UNASUR. Στις 30 Νοεμβρίου θα εγκριθεί το δεκαετές σχέδιο μέχρι το 2022-2024. Θα έχουμε το πρώτο μεγαλεπίβολο σχέδιο που Υπουργοί Υποδομών και Υπουργοί Ταξίας και Σχεδιασμού θα δώσουν το πράσινο φως σε μία πρόταση που σφυριλατείται εδώ και 10 χρόνια. Θα καταλήξει επιτέλους αυτή η προσπάθεια και θα ε, ε, χρηματοδοτήσουμε για 16 δισεκατομμύρια ευρώ 36 μακροσχέδια με συνεργασία ε, διαφόρων τοπικών τραπεζών αλλά αναζητώντας και στρατηγικούς εταίρους για αυτή την προσπάθεια επικοινωνίας για, αυτό το τεράσ... για αυτή την τεράστια πρόκληση της Λατινικής Αμερικής. Και επίσης θα έχουμε και συνεδρίαση των Υπουργών Επικοινωνιών της Γιουνασούρ για να εξετάσουν θέματα εκδημοκρατισμού, ε, βελτίωση της πρόσβασης στο διαδίκτυο, γιατί θα δημιουργηθεί ένα είδος δακτυλίου, ε, είδος δακτυλίου με επίκεντρο τη Βραζιλία. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα να δημιουργηθεί ένα τέτοιο δίκτυο. Είναι λοιπόν τεράστιο το δυναμικό της Λατινικής Αμερικής, αλλά εκρεμεί και το σημαντικό ζήτημα της εκρίζωσης της φτώχειας ή του περιορισμού των ανισοτήτων. Όσες προσπάθειες και αν κάναμε τα τελευταία χρόνια και όσες επιτυχίες και αν είχαμε, παρόλα αυτά το ζήτημα της φτώχειας και της ε, εξάλληψης των ανισοτήτων ε, εξακολουθεί να μας προβληματίζει. Και μάλιστα στη Λίμα τον Ιούλιο είχαμε την διακήρυξη κατά της ε, ανισότητας το θέμα της ε, υπέρβασης των ανισοτήτων είναι πολύ σημαντικό και σχετίζεται και με το ανθρώπινο κεφάλαιο, με την καινοτομία, με την τεχνολογία. δεν θα μπορέσουμε να συγκριθούμε με άλλες χώρες παρά την οικονομική ανάπτυξη που έχουμε αν δεν καταπολεμήσουμε προηγουμένως τεράστιες ανισότητες που διαπιστώνουμε στην περιοχή. Μία περιοχή σαν τη Λατινική Αμερική, σαν την Νότιο Αμερική, που είναι ενισχυμένη, ανανεωμένη στο πολιτικό διάνομο, με σταθερή μακροοικονομική ανάπτυξη, με σημαντικά αναπτυξιακά σχέδια και προγράμματα για την παιδεία, στα 8 συμβούλια, για θέματα υγείας, με κοινέ θέσεις σε πολυμερείς οργανώσεις. Θα πρέπει ε, να προσέξει ιδιαίτερα τη διαδικασία της ολοκλήρωσης. Σας ευχαριστώ πολύ και θα δώσουμε το παρόν στο Κίτο. Σας περιμένουμε γιατί η συμμαχία αυτή μεταξύ των κοινοβουλίων, αυτές οι σχέσεις είναι πολύ σημαντική πλατφόρμα για το κοινό μας μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Γενικέ. Θα ήθελα τώρα να αφήσουμε και λίγο χρόνο για συζήτηση, να δώσουμε το λόγο στους ευρωβουλευτές και τους βουλευτές. Παρακαλώ δύο λεπτά να μιλήσει ο καθένας και μετά η Γενική Γραμματέας θα μπορέσει να απαντήσει, να σχολιάσει τις διάφορες παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Το λόγο έχει ο κύριος Λουίς ε, Γιάννης. Ε, σου... Interesante. Ευχαριστώ την κυρία Γκλώρια Οκελή για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση και την κυρία Μεχία Βέλες για την ε, επίσης ενδιαφέρουσα ομιλία της. Το θέμα αυτό που μας απασχολεί, το θέμα των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής και, αυτό, και αυτή η κοινοβουλευτική συνέλευση Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής ε, είναι το κατεξοχήν πολιτικό κοινοβουλευτικό όργανο που βοηθά τις απρόσκοπτες σχέσεις μεταξύ των δύο υπήρων μέσω των ελεύθερα εκλεγμένων εκπροσώπων τους. Όπως είπε πριν από λίγο η Μπενίτα Φεραίρο, η Μπενίτα Φεραίρο είναι κατά κάποιο τρόπο η μητέρα αυτού του δημιουργήματος και στη διάσκεψη κορυφής του 2006. Δεν μιλάω μόνο για, για τη σύσταση του Ιδρύματος, είναι από ε, τους ιδρυτές ε, της ίδιας της ε, κοινοβουλευτικής συνέλευσης Eurolat από το 2006. Γιατί κάποιοι συνάδελφοι μου είπαν «Μα υπήρχε και προηγουμένως η Eurolat». Ναι, όντως υπήρχε. Προηγούμενα υπάρχουν πολλά και το γνωρίζει και ο Γινάσιος Αλαφράγκα. Αλλά συμπροέδρευε αυτό το προηγούμενο, το, τον πρόδρομο της Eurolat, αλλά το ποιοτικό άλμα που έγινε με αυτή την ε, νομική και πολιτική αναβάθμιση της ε, κοινοβουλευτικής συνέλευσης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην κυρία Μπενίτο. Γιατί βλέπουμε ότι σε κάθε συνεδρίαση υπάρχει μεγαλύτερη οριμότητα, μεγαλύτερη προσέλευση, καλύτερη ανταλλαγή απόψεων και μεγαλύτερη πρόοδος. Φυσικά δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος να κρίνω την πρόοδο της τελευταίας πενταετίας. Πάντως για όσους ε, δεν το γνωρίζουν, εγώ εκπροσωπώ εδώ την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι συντονιστής της ομάδας αυτής. Βέβαια έχουμε και άλλους ε, συναδέλφους και συντρόφους από την ομάδα, αλλά θα ήθελα να εκφράσω πραγματικά τη μεγάλη μου ικανοποίηση για τον τρόπο συνεργασίας ε, στην κοινοβουλευτική αυτή συνέλευση. Και θα ήθελα να πω κυρίω για του ε, Λατινοαμερικανού ε, ομολόγου μα. Μπορεί με να υπάρχουν ιδεολογικέ διαφορέ μεταξύ των Ευρωβουλευτών, μεταξύ του ΕΛΚ και των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ε, μεταξύ αυτών και των Πρασίνων ή της ΓΚΟΕ. Είναι 7 οι κοινοβουλευτικές ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά και οι 7 αυτές κοινοβουλευτικές ομάδες συμφωνούν παρόλο που δεν το έχουν γράψει πουθενά και δεν το έχουν δηλώσει επίσημα, έχουμε παρόμοιες απόψεις για τη Λατινική Αμερική, δηλαδή για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Λατινική Αμερική. Όλα τα πολιτικά κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι υπέρ της αναβάθμισης της σημασίας της Λατινικής Αμερικής στο πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πολλοί πιστεύουμε ότι η Λατινική Αμερική είναι η μεγάλη ξεχασμένη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο πρόγραμμά τη. Είδαμε από τα στοιχεία ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ούτε και εγώ το πιστεύω. Μερικέ φορέ μπορεί να λησμονείται από τα μέσα μαζική ενημέρωση, αλλά όλοι ξέρουμε ότι τα μέσα μαζική ενημέρωση δίνουν έμφαση στα προβλήματα, στι κρίσεις. Όταν υπάρχει πρόβλημα, όταν υπάρχει κρίση, τότε βρίσκεται αυτή η κρίση και στο επίκεντρο της προσοχής. Ε, βέβαια στο Κασμίρ έχουμε διαφιλονικία μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Ε, διεκδικείται και από τους δύο. Ε, φυσικά βρίσκεται το Κασμίρ στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής. Όταν όμως υπάρχει μια ομαλότητα της κατάστασης, ε, όπως και η ηρεμία, όπως στη Λατινική Αμερική τα τελευταία χρόνια, δεν απασχολεί αυτή η περιοχή την, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάνει και τη σημασία της για την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε σε πολιτικό επίπεδο είτε σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο. Και μάλιστα σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τη μετανάστευση, την ε, μετανάστευση της Λατινικής ε, Αμερικής προς την Ευρώπη, που με την οδηγία για τον επαναπατρισμό δημιουργήθηκε μια αποστροφή της Λατινικής Αμερικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση Εκεί που εξετάσαμε και επεξεργαστήκαμε το θέμα ήταν στην ομάδα εργασία για τη μετανάστευση της Eurolat. Και μάλιστα με τη σύσταση του παρατηρητηρίου δημιουργήσαμε μια καλύτερη αντίληψη και καλύτερη συνεννόηση για το θέμα αυτό. Νομίζω ήταν πολύ σημαντική συμβολή Τη ομάδα εργασία τη Eurolat. Θα δούμε βέβαια. σω αντιστραφούν οι τάσει και η μεταναστευτική ροή έχει τη φορά Ευρώπη Λατινική Αμερική και όχι την αντίστροφη που είχαμε στο παρελθόν. Αν συνεχιστεί κρίση στην Ευρώπη, οι μετανάστε έχουμε από την Ευρώπη προ τη Λατινική Αμερική. Εν πάση περιπτώσει... Συμφωνούμε για τα βασικά θέματα, εμπέδωση τη δημοκρατία, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο της παγκόσμιας τρομοκρατίας, ε, κρίζωση της φτώχειας, ισότητα των δύο φύλων, γιατί είναι κοινό προβληματισμός και για τις δύο υπήρους και εκεί υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες και θα πρέπει να επιτύρουμε τις προσπάθειες και είναι σωρία ε, ε, τα κοινά μας θέματα. Ένα άλλο ζήτημα που με ενδιαφέρει πολύ είναι το θέμα της ολοκλήρωσης. Εμείς είμαστε υπέρ της ολοκλήρωσης γιατί Είμαστε από την Ευρώπη και ευνοούμε την ολοκλήρωση παντού. Είμαστε υπέρ του Μερκοσούρ, τώρα έχουμε και το Γιουνασούρ. Η υποπεριφερειακή ολοκλήρωση στη Λατινική Αμερική είναι πολύ σημαντικό θέμα και μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι για σας σημαντικό σύμμαχος. Και έχουμε και το πλαίσιο ε, στρατηγικής συνεργασίας που ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει το πλαίσιο για το κοινό μας πεπρωμένο. Γιατί είχαμε ένα κοινό παρελθόν, σημεριζόμαστε συμμεριζόμαστε κοινέ αρχές και αξίες. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα μετατρέψουμε σε μια συνθήκη και για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σκουδέρο. Aquí ε. Σας ευχαριστώ κυρία Συμπρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γενική Γραμματέα της UNASUR για την παρουσία της και τη συμμετοχή της στην διάσκεψη αυτή της Eurolat. Έχω και εγώ κάποιες σκέψεις. Αναφέρθηκε στα μέσα της δεκαετίας, ε, μέσα σε τρία-τέσσερα χρόνια, η Κίνα θα εκτοπίσει την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ως στη θέση δεύτερου σημαντικού εμπορικού εταίρου της Λατινικής Αμερικής. Αυτό δείχνει τη δυσκολία που έχουμε στην ε, ενίσχυση των εμπορικών μας συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην εμφύση νέας πνοής. Έχουμε βέβαια το την πολιτιστική, κοινή πολιτιστική κληρονομιά, αλλά δεν αρκεί αυτό. Δεν αρκεί να χειρονόμαστε πίσω από την ε, πολιτιστική κληρονομία, γιατί φαίνεται ότι είναι πιο εύκολο για του Λατινοαμερικάνου να έχουν εμπορικέ συναλλαγές με την Κίνα από ό,τι με, τη από ό,τι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό φαίνεται γιατί σημειώνουμε, διαπιστώνουμε δυσκολίε στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Μερκοσούρ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαπιστώνουμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ακόμη την Λατινική Αμερική ως αποκλειστικό προμηθευτή πρώτων υλών. Αυτό το επιβεβαιώνει και η, ομιλία, η πρωινή ομιλία του Επιτρόπου Ταγιάννη. Γιατί είπε ο Επιτροπός ότι η Ευρώπη χρειάζεται συνεχή πρόσβαση στις πρώτες ύλες, κυρίως ε, ορυκτό και η ασυνέχεια στην πρόσβαση των πρώτων υλών δημιουργεί συγκρούσεις, είπε ο Επίτροπος. Δηλαδή υπάρχουν συγκρούσεις και πόλεμοι στον κόσμο όταν διαπιστώνεται μια συνέχεια στην πρόσβαση των πρώτων υλών. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση ε, για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής είναι πολύ πιο βαθιά και πολύ πιο ευρεία και δεν περιορίζεται μόνο στο εμπορικό σκέλος. Έχω την αίσθηση ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αρχίσει να αντιμετωπίζει ως ίσο, ισότιμο εταίρο την Λατινική Αμερική και την αντιμετωπίζει απλώς ως προμηθευτή πρώτων υλών, δεν πρόκειται να σημειώσουμε πρόοδο. Και σίγουρα η Κίνα και άλλες χώρες θα εκτοπίσουν σταδιακά την Ευρωπαϊκή Ένωση ως δεύτερο παγκόσμιο εμπορικό εταίρο της Λατινικής Αμερικής. Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, ένα μεγάλο τμήμα των επενδύσεων πάνε στην Καραϊβική, στους φορολογικούς παραδείσους της Καραϊβικής, βαθαίνοντας τις ανισότητες, οξύνοντας τους συστημικούς κινδύνους και δημιουργώντας προβλήματα ανισορροπίας και ανισότητας. Θεωρείται ότι ένα τρίτο τμήμα του παγκόσμιου πλούτου στον κόσμο βρίσκεται σε φορολογικούς παραδείσους, ε, αφορολόγητο δηλαδή, ενώ ταυτόχρονα σε... Χρειαζόμαστε φορολογικά έσοδα για να καλύψουμε τις ανισότητες μεταξύ των συμπολιτών μας και όχι φοροαπαλλαγές. Αυτά είναι μερικά από τα εμπόδια στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επαναλαμβάνω, η Λατινική Αμερική δεν είναι μόνο προμηθευτής πρώτων υλών. Αν υπάρξει μεταφορά τεχνολογίας και αν επιμείνουμε και στο θέμα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, γιατί λέμε μεταξύ των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που είναι συγκεντρωμένα σε ορισμένες χώρες και των θεμάτων της ασφάλειας φαίνεται ότι ο ανεπτυγμένος κόσμος εμποδίζει τον αναπτυσσόμενο ε, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη γνώση. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Αγκουστίν Διάς Δεμέρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να προλάβω την κυρία Φερέρο Βάλτνερ πριν φύγει και να κάνω κάποια σχόλια. Καταρχήν να συγχαρώ την κυρία Μεχία για την πολύ ενδιαφέρουσα και καλά τεκμηριωμένη και μεστή της ομίλια. Κυρία Φέρερο, καταρχήν συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο νέο Ίδρυμα, αλλά θα ήθελα να σας ε, παρακαλέσω για την προσοχή που χρειάζεται να δώσετε σε ό,τι αφορά την, μέχρι στιγμής, την ατελέσφορη ιδέα του παρατηρητηρίου των μεταναστευτικών ροών. Αυτή η ιδέα ήταν πολύ σημαντική και μάλιστα στην ομάδα εργασία, ο γερουσιαστή Πισαρόγιο και εγώ προσπαθούμε να προωθήσουμε αυτή την ιδέα του παρατηρητηρίου, αλλά θα πρέπει το παρατηρητήριο αυτό, αν όχι ως προς τη χρηματοδότηση, τουλάχιστον ως προς την ε, πολιτική υποστήριξη θα πρέπει να τύχει της στήριξης του Ιδρύματός σας. Δυστυχώς δεν άκουσα τίποτα από την κυρία Φέρερ Βάλνερ για τη μετανάστευση, τις μεταναστευτικές ροές. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική αρμοδιότητα αυτή για το Ίδρυμα και πιστεύω ότι αν την περιλάβετε στις αρμοδιότητες σας θα είναι πολύ σημαντικό. Ποια είναι λοιπόν, περιμένω μια αντίδραση, ένα σχολιασμό της πρότασης αυτής που έκανα από την κυρία Φέρερα Βαλνέρ. Καλώς τώρα να δώσω το λόγο στη Γενική Γραμματέα για να σχολιάσει τις πρώτες παρατηρήσεις και φυσικά να δώσω το λόγο και στην Πενίτα. Και θα έχουμε και δεύτερο ε, γύρο ομιλητών. Λάσαρο, Φιγκερέντο και Λουίς Σεράρια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τα λόγια του Λύση Γιάννης είναι πραγματικά αποκαλυπτικά και νομίζω ότι συνδυάζονται με αυτά που είπε και η κυρία Σκουδέρο. Όταν μιλούμε για την ε, υποπεριφερειακή ολοκλήρωση στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, διαπιστώνουμε ότι έχουμε σημειώσει πραγματικά εντυπωσιακή πρόοδο και είμαστε μία περιοχή του κόσμου που οι σχέσεις νότου-νότου, τα διδάγματα που αντλήσαμε και η πρόοδος που σημειώσαμε είναι εντυπωσιακά. Φυσικά μάθαμε και από τα παθήματά μας. Είχαμε υπερπληθωρισμό, είχαμε τη χαμένη δεκαετία, την προβληματική δεκαετία μεγάλες δυσκολίες και για τη δημοκρατία και για τις κοινέ μας αξίες αλλά φυσικά και για την οικονομία μας, την οικονομική μας κατάσταση. Αλλά ο σχετισμός δυνάμεων ε, έχει αλλάξει και ο τρόπος των σχέσεων έχει αλλάξει στη Λατινική Αμερική και εγώ είμαι αισιόδοξη γιατί πιστεύω ναι μεν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για την ε, Λατινική Αμερική και πιστεύει ότι είναι μεγάλο το πολιτικό της βάρος παρόλο που κάποιες στιγμές φαίνεται ότι αποσπάστηκε η προσοχή της προς άλλες από άλλες καταστάσεις όπως από την κρίση και φάνηκε αυτό και στο G20 γιατί και αναδυομένες οικονομίες όπως η Κίνα και η Ινδία στη τελευταία διάσκεψη κορυφής του G20 δεν είχαν σημαντικό μερίδιο στη συζήτηση ούτε οι αναπτυσσόμενες χώρες γιατί η συζήτηση σχεδόν μονοπολήθηκε στο G20 από την κρίση. Αυτό συμβαίνει μερικές φορές και με τη Λατινική Αμερική. Αυτό είναι κάτι προφανές. Πάντως, σίγουρα θα πρέπει να αλλάξουν οι σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα πρέπει να το αντιληφθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά θα πρέπει να βρούμε ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των διαφόρων φορέων. Η ΣΕΛΑΚ, για παράδειγμα, στις 3 Δεκεμβρίου θα εγκαινιαστεί η ΣΕΛΑΚ ως πολιτική ομπρέλα κατά κάποιο τρόπο Και είχαμε πρόσφατα τη Σύνοδο Κορυφής της Μποκοτά με τις πέντε χώρες που υπέγραψαν σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες. Θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να αναζητήσουμε το κοινό μας πεπρωμένο και σίγουρα η ενέργεια είναι ένας τομέας που θα βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής. Ο, η Βόρεια Χίλη έχει σημαντικά προβλήματα εφοδιασμού και οι υπόλοιποι των Άνδρων θα μπορούσαν να συνεργαστούν με τη Χίλη. Πάντως αυτό που βλέπω στους πολιτικούς μας και βλέπω και στα συμβούλια μας πώς αρχίζει και διαμορφώνεται ένα ε, ξεχωριστό δικό μας δόγμα. Και μάλιστα όσο ενισχύουμε τις εμπορικές συναλλαγές, τις διαπεριφερειακές, θα διαμορφωθεί και διαφορετική θέση μας ε, στην παγκόσμια σκηνή. Και φυσικά περιφερειακή ολοκλήρωση θα συμβάλλει σημαντικά σε αυτή την αλλαγή της πολιτικής μας παρουσίας στον κόσμο. Η Μπένιτα τώρα. Θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε, με την άδειά σας, να ευχαριστήσω θερμότατα τους ομιλητές και να σχολιάσω αυτό που είπατε. Ε, Έψεχνα το καταστατικό του Ιδρύματος και στο άρθρο 2 εδάφιο 2 στους στόχους του Ιδρύματος ε, αναφέρεται ρητά και η μετανάστευση. Αυτό που διαβάζω όμως είναι ότι πρόκειται για τις δραστηριότητες ε, που επισημαίνουν στις διασκέψεις κορυφής οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και αυτοί επισημαίνουν τους προσανατολισμούς και τις προτεραιότητες. Βρισκόμαστε σε μια προκατακτική φάση. Ακόμη βρίσκεται στα σπάργανα ουσιαστικά αυτό το Ίδρυμα και ακόμη το γαλουχούμε. Είναι σε βάση θυλασμού και μάλιστα δεν έχουμε αρκετό γάλα για να τροφοδοτήσουμε αυτή τη στιγμή το έμβριο αυτό, το, όχι το έμβριο, μάλλον το νήπιο, το βρέφος αυτό που είναι το Ίδρυμα. Θα συνεχίσει όμως να μεγαλώνει το Ίδρυμα αυτό και να συμβάλλει και στη διάσκεψη κορυφής του Σαντιάγο στη Χιλή. Πάντως, όσο εμπεδώνεται και κατοχυρώνεται η θέση του Ιδρύματος, τόσο θα περιλαμβάνει και περισσότερα θέματα. Γιατί, από ό,τι ξέρω, υπάρχει και μια ειδική επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ασχολείται με το θέμα αυτό. Οπότε, μας ενδιαφέρουν τα συμπεράσματα των εργασιών σας και μαζί με τον Χόρχε Βαλντές θα δούμε πώς μπορούμε να τα λάβουμε υπόψη. Όλα τα θέματα είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν μπορώ να αναλάβω επίσημη δέσμευση γιατί ακριβώ βρισκόμαστε σε πολύ προκατακτική φάση. Ευχαριστώ. Ε, η μητέρα του Ιδρύματος είναι πολύ σημαντική. Η μάνα πάντα βρίσκει τρόπο. Έχουμε εμπιστοσύνη λοιπόν στο ένστικτο της μάνας για το μέλλον του παιδιού. Η Σιμένα Βιδά Λάσαρο. Σας ευχαριστώ. Είμαι βουλευτής από την Χιλή σε ό,τι αφορά τη μαμά να αποτίσω φόρο τιμής και στην κυρία Μπατσελέ την πρόοδό μας που είναι ε, πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών στα Ηνωμένα Έθνη. Θα ήθελα να απευθύνω χαιρετισμό προς την Κοινοβουλευτική Συνέλευση ε, και στην ε, Γενική Γραμματέα της Ουνασούρ. Μιλήσατε για τις μεταρρυθμίσεις του κράτους, για τη μεταμόρφωση του κράτους και για το έργο της Γιουνασούρ. Έχω ένα σχόλιο παρόμοιο με τις ε, γερουσιαστού του. Σίγουρα έχουμε πρόθεση ολοκλήρωσης, αλλά σε ό,τι αφορά τους φυσικούς πόρους μας, ο φόβος των εκπροσώπων μας είναι η α, απώλεια των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών μας αγαθών. Έχουμε λοιπόν την κοινωνική πίεση απέναντι στους διάφορους οικονομικούς δείκτες. Έχουμε βέβαια μια θετική μακροοικονομική ανάπτυξη και έχουμε υψηλά ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης, αλλά όπως ακούσαμε το πρωί και το γνωρίζουμε και εμείς, υπάρχουν τεράστιες ανισότητες ακόμη στη Λατινική Αμερική και αυτό το ζήτημα πρώτα απ' όλα θα πρέπει να επιλύσουμε. Εμένα με απασχολεί την αντισυστημική κινητοποίηση που διαπιστώσαμε και ε, Είδαμε και το κίνημα των αγανακτισμένων και υπάρχουν διάφορα τέτοια κινήματα κατά της παγκοσμιοποίησης. Έχουμε δύο στρατόπεδα. Μερικοί που θέλουν να διαφυλάξουν ε, το κεκτημένο τους και την ευημερία και άλλοι που θέλουν να την ε, ε, ανακτήσουν ή να έχουν πρώτη πρόσβαση σε αυτή την ευημερία. Το θέμα είναι πώς θα προωθήσουμε αφενός την ολοκλήρωση και τη συνεργασία, αντιμετωπίζοντας όμως και τους κόδωνες του κινδύνου για τη μεταρρύθμιση του κράτους και την τροποποίηση ή την ε, κατοχήρωση του αναπτυξιακού μας μοντέλου. Τι συνέβη στο Γιούνασουρ, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ το λόγο κυρία Ήλντα Φιγκερέντο. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να χαιρετήσω και εγώ τη Γενική Γραμματέα της Γιονασούρ, αλλά και όλους τους βουλευτές, άνδρες και γυναίκες, που συμμετέχουν σε αυτή την κοινοβουλευτική συνέλευση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε υποδεχόμαστε με χαρά τους συναδέλφους της Λατινικής Αμερικής. Ακούσαμε πολλά θέματα στην πρωινή συζήτηση. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ σε λίγα σχόλια και να σας εκθέσω τη θέση μας. Οι ανησυχίες που έχουμε σήμερα με την σημερινή κρίση, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια κρίση που οξύνεται σε πολλές χώρες, όπως στη δική μου πατρίδα την Πορτογαλία, για παράδειγμα, τη, τη βδομάδα αυτή στην Πορτογαλία, την Πέμπτη η στις 24 του μηνός, θα πραγματοποιηθεί γενική απεργία των εργαζομένων, γιατί πραγματικά έχουμε μια ένα σύμφωνο ύφεση, ένα σύμφωνο επίθεση κατά των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η οικονομία μας είναι πολύ ευάλωτη η κατάσταση πολύ χαλεπή, αλλά γίνεται μια ε, επίθεση κατά των δικαιωμάτων των εργαζομένων, κατά των δικαιωμάτων των πολιτών, κάτι που μας δημιουργεί μια τεράστια κοινωνική παλιδρόμηση. Μας προβληματίζει λοιπόν σοβαρότατα και μας θορυβεί αυτή η κατάσταση, όχι μόνο στην Πορτογαλία και άλλο γνωρίζουμε την κατάσταση στην Ελλάδα, αλλά βλέπετε ότι και σε άλλες χώρες μετατοπίζεται η κρίση, στην Ιταλία, στην Ισπανία και το καθεξής. Με πολύ μεγάλη ανησυχία λοιπόν παρατηρούμε αυτή την κατάσταση με μια απορρίθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, με πραγματική δικτατορία των αγορών εις βάρος της δημοκρατίας. Η δημοκρατία φαίνεται ότι αποδυναμώνεται και κλονίζεται όλο και περισσότερο στις διάφορες χώρες που μαστίζονται από την κρίση και είναι οξύτατες και οι ανησυχίες στον κοινωνικό τομέα. Η Πορτογαλία ήδη βρίσκεται σε ύφεση, η φτώχεια επιδεινώνεται, η ανεργία ενισχύεται και οι κοινωνικές ανισότητες επίσης οξύνονται. Παρ' όλα αυτά οι μεγάλες επιχειρήσεις εξακολουθούν να έχουν υπέρογκα κέρδη, οι φορολογική παράδεισοι να ανθούν, ενώ ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού να χάνει τη δουλειά του και να βλέπει το εισόδημά του να εξαφανίζεται. Αυτή η κατάσταση είναι νεοφανής, πολύ ανησυχητική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη σε όλες αυτές τις αναλύσεις που κάνουμε ε, Αποκινούμε τη Eurolat. Η, θέση μας είναι πολύ επικριτική απέναντι σε ορισμένες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου που συνάπτονται με χώρες Λατινικής Αμερικής. Για παράδειγμα, η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με την Κολομβία ή το Περού δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Εμείς θέλουμε να ενισχυθεί μεν η συνεργασία με τις χώρες Λατινικής Αμερικής, αλλά με ισότιμο τρόπο, με σεβασμό των, εργα... των δικαιωμάτων των εργαζομένων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε οι εργαζόμενοι αυτοί είναι Ευρωπαίοι υπήκοοι είτε είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. Αλλά θέλουμε και στις χώρες Λατινικής Αμερικής να γίνονται σεβαστά και τα δικαιώματα των εργαζομένων και η φυσική πόροι και η κοινωνική πρόνοια. Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω όλα αυτά τα σημεία. Δεν είμαστε κατά του εμπορίου μεταξύ των δύο όχθεων του Ατλαντικού, αλλά θέλουμε να γίνεται με ισότιμο τρόπο και όχι εις βάρος των δικαιωμάτων και για να βελτιώσουμε τις βιωτικές συνθήκες των συμπολιτών μας και όχι για να βελτιώσουμε μόνο το κέρδος των πολυεθνικών γιατί συνεχίζουν οι πολυεθνικές ε, να συσσωρεύουν κέρδη εις βάρος των εργαζομένων και των λαών. Σε ό,τι αφορά την μετανάστευση, πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αλλάξει θέση απέναντι στη μετανάστευση. Εμείς ταχθήκαμε στην ΚΟΕ και Σκανδιναβική Αριστερά κατά της οδηγίας ε, τις οδηγίες επαναπατρισμού ή τις οδηγίες του ονίδους όπως την αποκαλούσαμε. Θέλουμε να αναθεωρηθεί η οδηγία αυτή και να λάβει υπόψη τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων και των Ευρωπαίων και των εξοκοινωτικών. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μια ισοτιμία των δικαιωμάτων και των καταστάσεων. Ένα θερμό χαιρετισμό επίσης θέλω να σας απευθύνω. Είμαστε μαζί σας για να συνεχίσουμε το έργο μας και να ενισχύσουμε την συνεργασία μεταξύ μας γιατί πιστεύουμε ότι είναι σημαντική. Τώρα έχουμε τον βουλευτή Ροντρίγκο Καμπέσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Συμπροεδρεύουσα. Θα ήθελα εκ μέρους και του κόμματός μου να ευχαριστήσω την δόκτωρα Μαρία Μαχία για τη θαυμασία παρουσίασή της. Θα και ήθελα να προσθέσω το εξής. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τους Λατινοαμερικάνους. Η πρόκληση στον 21ο αιώνα είναι η πολιτική και η οικονομική και η κοινωνική ενσωμάτωση, η ολοκλήρωση. Η λύση των προβλημάτων μας δεν θα βρεθεί ούτε από την Ευρώπη ούτε από την Αφρική, είναι στα χέρια μας. Έχουμε μια δυναμική ολοκλήρωση που έχει ξεκινήσει στην αρχή του 21ου αιώνα και αυτό είναι κάτι τελείως καινούριο στην ιστορία μας. Το όνειρό μας είναι η Λατινική Αμερική να γίνει ένα νέο οικονομικός συνασπισμός στο σύνολο των εθνών. Θα θέλαμε η ενίσχυση αυτή της Λατινικής Αμερικής να μην είναι πολιτικής χρειάς ούτε και κομματικής. Ε, θέλουμε να είναι μία ανταπόκριση στις σημερινές οικονομικές εξελίξεις. Λοιπόν, θα θέλαμε πολύ να φέρουμε τη Λατινική Αμερική να καταφέρουμε η Λατινική Αμερική να ξεπεράσει αυτή την κρίση. Πιστεύουμε ότι σε μία δεκαετία ακόμη ο καπιταλιστικός κόσμος θα πρέπει να βρει λύσεις για αυτές τις φούσκες που εκρήγνυνται κατά τρόπο χρόνιο, θα έλεγα, και κρίσιμο. Ε, υποστηρίζουμε αξίες όπως ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, και ακόμη πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να ανταγωνιζόμαστε αλλά να συνεργαζόμαστε όσον αφορά τις βιομηχανίες μας και τις παραγωγές μας. Πρέπει να χρηματοδοτήσουμε την ανάπτυξή μας, να χρησιμοποιήσουμε τις οικονομίες για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε την πολιτική μας, κοινωνική μας, οικονομική μας ανάπτυξη. Η Μαρία Μαχία είπε ότι τελικά είναι εφικτό μια πολιτική και κοινωνική ομάδα να μπορέσει να ενωθεί για την ειρήνη σαν παγκόσμια αξία. Η σχέση μας όμως με διάφορα μέρη του κόσμου όπως ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει ακριβώς να ρίζεται σε αυτές τις αξίες. Υπάρχει κάτι ακόμη που θα ήθελα να πω. Η διαδικασία της ολοκλήρωσης που ακολουθούμε, η διαργασία αυτή ε, και αυτό είναι κάτι που δεν αναφέρθηκε από την κυρία Μαχία. Έχει ως εξή. δηλαδή δεν ανησυχούμε μόνο για ε, τα ωραία λόγια γύρω από την ολοκλήρωση. Θα θέλαμε περισσότερο να εξετάσουμε τα προβλήματα και τους τομείς ε, που θα θυγούν καθώς προχωράμε προς την ολοκλήρωση. Έχουμε Έχουμε τώρα μία τράπεζα ανάπτυξης Λατινικής Αμερικής. 20 ε, δις είναι το κεφάλαιο και πολλές λατινοαμερικές χώρες έχουν προσχωρήσει, δεν έχουν ακόμη ενεργοποιήσει όλες τη σχετική νομοθεσία, αλλά είναι μια νέα δομή και θα είναι έτσι δυνατόν να έχουμε χρηματοδότηση της ανάπτυξης μέσω αυτής της τράπεζας και αυτό θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τις εμπειρίες που είχαμε εμείς με την Παγκόσμια Τράπεζα. Η Παγκόσμια Τράπεζα προσδιορίζει τις οικονομικές πολιτικές που πρέπει να ακολουθηθούν προτού χρηματοδοτήσει. Αυτό βεβαίως επέδρασε στην παιδεία και στην υγεία ε, όσον αφορά τις χώρες που έλαβαν τέτοια χρηματοδότηση για την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική. Ε, έχουμε τη ρύθμιση Πέτρο Καρύμπε βεβαίως και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τους εαυτούς μας σαν σημαντικός παραγωγός ε, πετρελαίου, ραφιναρισμένου και αργού και με τον τρόπο αυτό ε, πρέπει να διασφαλίσουμε την ενεργειακή μας επάρκεια, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Αυτή είναι μια κατεύθυνση σημαντική, όπως ήδη έχει αναφερθεί. Ακόμη, έχουμε ένα πρότυπο ενδεχόμενου νομίσματος, το Σούκρε, ε, Βενεζουέλα, Κούβα, Νικαράγουα κτλ ενδέχεται να συμμετάσχουν για τις εμπορικές συναλλαγές τους. Δεν χρησιμοποιούμε δηλαδή το δολάριο ούτε το ευρώ, χρησιμοποιούμε το δικό μας νόμισμα, το θεωρητικό για τις εμπορικές μας συναλλαγές. Παρόμοια αρρύθμιση υπάρχει και στο Μερκοσούρ, αλλά το Σούκρε που κάποτε έμοιαζε να είναι ουτοπία, πριν δημιουργηθεί το ευρώ, παρόλα αυτά το Σούκρε εξακολουθεί να λειτουργεί και ε, θα μπορούσε να εξελιχθεί και να καλύψει όλη τη Λατινική Αμερική σαν εμπορικό νόμισμα για εμπορικές συναλλαγές. Ο Γενικός Διευθυντής της Γιούλα που μίλησε σήμερα το πρωί είπε ότι ένα από τα πιο, μία από τις πιο σημαντικές απειλές ήταν η επανιδιωτικοποίηση της οικονομίας μας. Βεβαίως, όλοι μας έχουμε μία, ένα όραμα και δεν συμφωνούμε με τους Ευρωπαίους που θεωρούν ότι το πεπρωμένο της Λατινικής Αμερικής είναι ένα πολύ μόνο πρωτεσίλες. Πιστεύουμε ότι το διαπεριφερειακό εμπόριο είναι ο σωστός δρόμος. Έχουμε και μία πρόκληση τεχνολογική και πιστεύουμε ακόμη ότι οι εξαγωγικές μας πλατφόρμες θα μας δώσουν πρόσβαση πιο προοδευτική στις αγορές. Ο κύριος Πισάρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ και για τις ομιλίες και για τις πολύ εύστοιχες παρατηρήσεις που ακούσαμε όλο το πρωί σήμερα αλλά και χθες ολόκληρη την ημέρα. Αναμφίβολα ε, από το πρίσμα της Λατινικής Αμερικής η βλέψη αυτή προς την ολοκλήρωση είναι ο σημαντικότερος μας στόχος και αυτό το επισημαίνουμε σε όλες τις ευκαιρίες που έχουμε ως βουλευτές Προσπαθούμε να συγκεκριμενοποιήσουμε τους διάφορους μηχανισμούς και επίπεδα ολοκλήρωσης στην Λατινική Αμερική. Και από αυτή την άποψη η εμπειρία στη UNASUR, στην Ένωση Νοτιοαμερικανικών Εθνών, ήταν μια πολύ θετική εμπειρία. Ναι, μεν είχαμε δυσκολίες και προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα αξιοποιήσαμε διάφορες ευκαιρίες και συνεχίσαμε αυτή την πορεία της ολοκλήρωσης. Θα ήθελα να εκφράσω μια επιφύλαξη, ε, ευκαιρία και της παρουσίας σας κυρία Γενική Γραμματέα. Οι αποφάσεις που υιοθετούν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ή οι πρωτοβουλίες των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων θα πρέπει κάποιος να τις εφαρμόσει για να έχουν νόημα. Κάποιος, κάποιες φορές θα πρέπει να τις εκτελέσει. Αλλιώς θα μείνουν σε επίπεδο ε, διακήρυξης προθέσεων. Αν δεν μεταφέρουν μετασαρκωθούν, αν δεν αποκτήσουν σάρκα και οστά, δεν έχει νόημα απλώς ε, να εκφράζουμε αγαθές προθέσεις και μετά να τις αφήνουμε ανεφάρμοστες. Το λέω αυτό γιατί κάποια στιγμή ο πρόεδρος Λούλα και άλλοι πρόεδροι είπαν ότι ε, η Γιούνα Σούρη έπρεπε να έχει και μια κοινοβουλευτική συνιστόσα και ε, έλαβαν την απόφαση να δημιουργήσουν και μια κοινοβουλευτική ε, πτυχή στη Σούρ. Αυτή όμως την απόφαση την έλαβαν οι πρόεδροι. Δεν συμμετείχαν τα κοινοβούλια και δεν ξέρουμε ποιο θα είναι ο ρόλο αυτού του κοινοβουλευτικού βραχίωνα τη Σούρ. Θα είναι ελεκτικό ο ρόλο, ε, ε εκτελεστικό, τι αρμοδιότητε θα έχει, τι πεδίο εφαρμογή θα έχει. Είναι πολύ ε, λεπτό αυτό το θέμα. Και επειδή υπάρχει και επικάλυψη με, άλλ, με άλλες κοινοβουλευτικές οργανώσεις, δημιουργείται ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα για το τι χαρακτήρα θα έχει αυτή η κοινοβουλευτική συνιστόσα της Γιουνασούρ. Επίσης, οι πρόεδροι επιρρύπτουν τις ευθύνε σε συγκεκριμένη χώρα, σε συγκεκριμένο πρωθυπουργό ή πρόεδρο, κάτι που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση. Γιατί είχαμε χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας πολύ θετικής πρωτοβουλίας που έμεινε ανεφάρμοστη στην πράξη γιατί δεν έχει την υποστήριξη των κοινοβουλίων, οπότε έμεινε τελικά στα χαρτιά. Είχαμε βέβαια τον Αντιπρόεδρο Καρσία Λινέρα της Βολιβίας σε μια συνεδρίαση που δεν είχε επιτυχία γιατί τα ίδια τα κοινοβούλια στις διάφορες προσπάθειες που έκαναν δεν υποστήριξαν αυτή την πρωτοβουλία. Πιστεύω ότι η Γενική Γραμματέας της UNASUR θα πρέπει ε, να συμφωνήσει για τον τρόπο λειτουργίας αυτής της κοινοβουλευτικής πλατφόρμας με τρόπο που να συνάδει με, με τις φιλοδοξίες της UNASUR και να συμπληρώνει τις τα υπόλοιπα επίπεδα της ε, Μερκοσούρ, της Λατινοαμερικανικής ε, Συνέλευσης, της Συνέλευσης των Άνδεων, γιατί υπάρχουν διάφορα κοινοβουλευτικά φόρα. Και αυτό το λέω γιατί πρόσφατα ανέκυψε το θέμα της κοινοβουλευτικής συνιστώσης της Σούρ. Ένα άλλο θέμα άπτεται της ερώτησης του κυρίου Διασδεμέρο προς την πρόεδρο του Ιδρύματος ε, Γιούλακ, κυρία Μπένιτα Φερέρα. Μπένιτα, αν οι πρόεδροι τη συνόδους κορυφής εγκρίνουν τις δικές μας προτάσεις και αποφασίσουν να δεχτούν την πρότασή μας για τη σύσταση παρατηρητηρίου για των μεταναστευτικών ροών, εμείς θεωρήσαμε ότι εν μέρει ήταν ευθύνη και του Ιδρύματος να ε, εφαρμόσει αυτή την πρόταση του παρατηρητηρίου με την πολιτική υποστήριξη φυσικά των αρχικών κρατών και κυβερνήσεων αλλά και της κοινοβουλευτικής συνέλευσης. Αυτή ήταν η δική μας αντίληψη για την εντολή στην οποία συμμετέχουμε, στις επιτροπή στην οποία συμμετέχει και ο κύριος Δίας Δεμέρα και εμείς. Είχαμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για τον τρόπο λειτουργίας του παρατηρητηρίου, για το στόχο του παρατηρητηρίου, για τη μορφή που θα πρέπει να έχει, για την αποστολή του παρατηρητηρίου και θέλουμε το συντομότερο δυνατό να καταλήξουμε σε μια οριστική πρόταση. Αύριο γίνεται. Αυτό που θα σας ζητούσε λοιπόν, γνωρίζοντας και το χαρακτήρα σας, πιστεύω ότι η ανάπτυξη αυτού του βρέφους θα είναι πραγματικά ε, εντυπωσιακή. Γιατί θέλουμε το συντομότερο δυνατόν να μεγαλώσει αυτό το βιονικό κατά τη γνώμη μου βρέφος μια και θα έχει τέτοια μάνα, τέτοια μητέρα σαν και εσάς. Όταν πριν από λίγα χρόνια προσπαθήσαμε να δώσουμε σάρκα και οστά στο παρατηρητήριο για τη μετανάστευση, μας είπαμε περιμένετε πρώτα το Ίδρυμα, γιατί το Ίδρυμα θα είναι ο κατάλληλος φορέας για να ε, δώσει σάρκα και οστά στην πρωτοβουλία για το παρατηρητήριο. Θα πρέπει ήδη από τώρα όμως να υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση, γιατί υπάρχει μια πολιτική δέσμευση που ε, χρειάστηκε πολύ καιρό και πόδινες διαπραγματεύσεις για να την υλοποιήσουμε και υπήρχε μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τα μεταναστευτικά ζητήματα και νομίζω ότι το παρατηρητήριο είναι καλύτερο, το καλύτερο φόρουμ για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες τριβές. Θέλουμε να μετατραπεί το θέμα της μετανάστευσης σε ευκαιρία γιατί δεδομένων των εξελίξεων που είχαμε σε θέματα μετανάστευση μεταξύ των δύο εταίρων, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή τώρα να προωθήσουμε το παρατηρητήριο. Φαντάζομαι ότι αύριο στην Επιτροπή και ο Ντίας Δεμέρα και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής θα εγκρίνουμε την οριστική απόφαση για τη σύσταση του παρατηρίου με πολύ συγκεκριμένη πρόταση και ελπίζουμε το συντομότερο δυνατό σε μια συνεδρίαση εργασίας να κάνουμε όλα τα απαραίτητα ώστε να εφοδιάσουμε το μωρό με το γάλα που χρειάζεται. Νομίζω ότι αυτό είναι κοινό στόχο για όλου. Ευχαριστώ. Και τελευταία παρέμβαση του κυρίου Έντουαρτ Κοσούσνικ. Σα είπα ότι έχουμε ελάχιστο χρόνο και θέλουμε να ακούσουμε και τα τελικά σχόλια. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και σας συγχαίρω για την σωστή προφορά του ονόματός μου. Uh, Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους uh, συναδέλφους, τους ομολόγους μας από τις Λατινοαμερικανικές uh, βουλές. Θα ήθελα να σας μεταφέρω το χαιρετισμό και την εμπειρία όχι μόνο της πατρίδα μου της Τσεχίας, αλλά και των άλλων χωρών που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Παρακαλώ λίγη ησυχία, λέει ο Πρόεδρος, γιατί δεν ακούμε τον ομιλητή. Εμείς είμαστε λίγο μεγαλύτεροι από τη Eurolat, γιατί αν δεν κάνω λάθος η Eurolat ε, ιδρύθηκε το 2006 και εμείς μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, αλλά έχουμε λίγο μεγαλύτερη πείρα. Κατά τη γνώμη μας είναι σημαντική αυτή η πλατφόρμα της Eurolat για να συζητούμε όχι μόνο θέματα εμπορικών συναλλαγών, αλλά και μεταναστευτικά ζητήματα, θέματα αλληλεγγύης, αλλά και άλλα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ των δύο εταίρων. Ίσως ε, να φαίνεται ότι η χώρα, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Λιθουανία ε, ενδιαφέρονται λιγότερο για τη Λατινική Αμερική από ότι χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι σωστή και ακριβής αυτή η εντύπωση. Γιατί η εμπειρία μας από τις νέες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, η εμπειρία μας από την ολοκλήρωση είναι πολύ θετική και οι συνάδελφοι που με γνωρίζουν ξέρουν ότι ανήκω στην ε, ομάδα των μεταρρυθμιστών και συντηρητικών. Οπότε θα μου πούν αυτά που λες δεν συνάδουν με τη γενική θέση της ομάδας σου. Πάντως πιστεύω ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο υπήρων είναι πολύ σημαντική γιατί ο κόσμος γίνεται όλο και πιο μικρός. Γι' αυτό και πρέπει να αναζητήσουμε φίλους. Και νομίζω ότι η φιλία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να φανταστούμε. Σε ό,τι αφορά το παρατηρητήριο για τις μεταναστευτικές ροές και στις νέες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα νέο φαινόμενο που αντιμετωπίζουμε είναι το εξής. Στην Πράγα, η κοινότητα των Ισπανοφώνων ε, αυξήθηκε σιτά τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει έντονη μεταναστευτική ροή από τη Λατινική Αμερική προς α, ακόμη και τις νέες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην μιλάμε μόνο για εμπόριο και πρώτες ύλες, να, μιλάμε, να μιλήσουμε και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να μιλήσουμε και για την ελληνική και γι' αυτό χρειαζόμαστε το παρατηρητήριο μεταναστευτικών ροών. Γιατί αν υπάρχουν μετανάστες θα πρέπει να τους προστατεύσουμε, να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματά τους όποια φορά και αν έχουν αυτές οι μεταναστευτικές ροές. Εγώ είμαι υπέρ της ίδρυσης του παρατηρητηρίου για τις μεταναστευτικές ροές. Είμαι ενθουσιώδης υπέρμαχος αυτής της πρότασης. Ευχαριστώ το λόγο και γενικοί γραμματές. Ευχαριστώ για τα ελάχιστα λεπτά που μου δίνετε στο τέλος για να ολοκληρώσω. Και να ευχαριστήσω θερμά όλου του ευρωβουλευτέ και του βουλευτέ των χωρών τη Λατίνική Αμερική για τη συμμετοχή του στη συζήτηση. Νομίζω ότι μπροστά μα έχουμε μακρύτατο δρόμο και όπω είπε και ο Ευρωβουλευτής Κοτσούσνικ, Έντουαρτ, Έντουαρτ. Ο κόσμος ε, γίνεται όλο και πιο μικρός, γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρχει αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη. Και αυτό εμπόδισε την ολοκλήρωση στο Μερκοσούρ. Υπήρχαν μεγάλες διαφορές μεταξύ μας. Δεν ε, γνωριζόμασταν ουσιαστικά μεταξύ μας, παρόλο που ήμασταν γειτονικέ χώρες δεν είχαμε συζητήσει ε, ποιο μπορεί να είναι το κοινό μας αναπτυξιακό μοντέλο και το κοινό μας μέλλον. Δεν υπήρχε τέτοια επιθυμία συζήτησης προηγουμένως. Τώρα όμως υπάρχει. Και αυτή η συζήτηση πια είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα της Ήπειρου. Γιατί όντως υπάρχει, υπάρχουν αγανακτισμένοι και στη Χιλή και στην Κολομβία. Θα γίνει στις 24 του μηνός ε, ε, παναμερικανικό συλλαλητήριο και στη Χιλή έχουμε, θα έχουμε διαδηλώσεις και των ε, ε, φοιτητών και των εργαζομένων γιατί ξοδέψαμε τόση ενέργεια για να καταρτήσουμε και να σπουδάσουμε φοιτητές και βλέπουμε ότι αυτοί οι φοιτητές ε, αποφοιτούν και δεν έχουν δουλειά και είναι λογικό να είναι αγανακτισμένοι και να διαμαρτύρονται. Θα πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, να μεγαλώσουμε ε, την μέση τάξη, τη μεσαία τάξη, γιατί όπως είπε η Κίλντα, είναι δεινή η κατάσταση που αντιμετωπίζουν πολλοί εργαζόμενοι. Έχουμε πια και νέους από πανεπιστημίων που δεν μπορούν να βρουν μια θέση εργασίας. Αυτό είναι ένα κοινό πρόβλημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Λατινική Αμερική και εντάσσεται στις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και γνωρίζω ότι οι πρόεδροι το έλαβαν αυτό υπόψη και, και τα κοινοβούλια το ίδιο και ο αντιπρόεδρος της Βολιβίας έκανε μια προσπάθεια για την συνεδρίαση αυτή που τελικά πέτυχε αλλά και ο πρόεδρος της Βουλής του η σημερινή κάνουμε μια νέα προσπάθεια για να δούμε τι μορφή θα μπορούσε να έχει αυτό το νέο κοινοβούλιο της Γιούνασουρ τι μορφή θα δώσουμε σε αυτή την κοινοβουλευτική διάσταση. Με συνεργασία όμως των βουλευτών και πιστεύω ότι το Φεβρουάριο στον Ισημερινό θα σημειωθεί μια πρόοδος, θα γίνει μια καλή συζήτηση, γιατί θέλουμε μια και ολοκλήρωση και των κοινοβουλίων. Και το είπαμε αυτό και στην Κοτσαμπάμπα. Η Γιουνασούρ είναι σημαντική, αλλά σημαντική Ένωση νοτιοαμερικανικών εθνών δεν νοείται χωρίς ε, ένωση των κοινοβουλίων. Γιατί έχουμε διάφορες κοινοβουλευτικές ε, οργανώσεις του Μερκοσούρ, του, των Άνδεων, αλλά θα δούμε πώς θα προβλέψουμε κάτι αντίστοιχο και για τη UNASUR. Και το πλεονέκτημα της UNASUR είναι ότι οι υπουργοί των εκτελεστικών κλάδων πραγματικά ε, έχουν εκτελεστική εξουσία και μπορούν να εφαρμόσουν και εμπράκτο τι αποφάσεις που λαμβάνουν. Δεν μένουν μόνο στα χαρτιά. Και μάλιστα την Παρασκευή οι Υπουργοί ε, Εθνική Οικονομίας και Οικονομικών που θα ασχοληθούν με το θέμα της Τράπεζας του Νότου, γιατί η Ουρουά είναι η πέμπτη χώρα που θα θέσει σε εφαρμογή αυτό το σχέδιο. Ήδη το ενέκρινε η Γερουσία και πριν τη 15η Δεκεμβρίου θα περάσει και στην Βουλή ώστε να τεθεί σε εφαρμογή. Αυτό που χρειάζεται είναι τόλμη και θάρρος και η, Νότια, Αμερική, η Νότια Αμερική δείχνει ότι με θαραλέα μέτρα, ε, γιατί έχουμε το... Αναφέρθηκε το σχόλιο και τι θα γίνει με την Τράπεζα του Νότου, ποιος θα τη διαχειριστεί, ποιος θα τη διοικεί. Όμως χρειαζόμαστε αυτά τα θαραλέα μέτρα, αυτά τα τολμηρά μέτρα, γιατί μας χρειάζεται για την ολοκλήρωση αυτό το νέο αρχιτεκτόνημα. Και έχουμε πραγματικά μεγάλες ευκαιρίες και δυναμικό για να επιδιώξουμε ολοκλήρωση και μεταξύ μας, αλλά και να βελτιώσουμε τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους θερμά. συγκινήθηκα πραγματικά με τις παρεμβάσεις με τις δεσμεύσεις σας και την προσήλωσή σας. Γιατί πιστεύω ότι αυτή η κοινοβουλευτική συνέλευση Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής δίνει σημαντική όθηση και αν ε, ένα τμήμα του ενθουσιασμού σας ε, το συμμεριστούν και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα δείξουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για να προωθήσουν αυτή τη σημαντική συμμαχία και μάλιστα σε περίοδο κρίσης. Ευχαριστώ. Vamos a, a dar las gracias. ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά τους ε, θαυμάσιους ε, διερμηνείς. Τους ευχαριστούμε θερμά για την καλοσύνη που είχαν να ε, ε, ξεπεράσουν και το ωράριό τους και να παραμείνουν ακόμα λίγο στη συνεδρίαση. Και για τα πραγματικά καταληκτικά σχόλια, κυρία Μπενίτα Φερερό. Σας ευχαριστώ κυρία Συμπρόεδρε. Κύριε Γερουσιαστά, το μήνυμα και το δικό σας και του Ευρωβουλευτού Διέσδε Μέρα. Όπως είπα και προηγουμένως, βρισκόμαστε στα σπάργανα του Ιδρύματος. Οι στόχοι μας είναι πολλοί και είμαι πρόθυμη για διάλογο μαζί σας. Όταν οριστικοποιηθεί το σχέδιό σας θα το συζητήσουμε, θα βρεθούμε και θα το εξετάσουμε και κατόπιν θα δούμε πώς ε, θα το εντάξουμε στους στόχους μας γιατί δεν υπάρχει ρητά στους στόχους αυτό. Αλλά για κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε και συνεισφορές και κονδύλια, γιατί προς το παρόν το ταμείο είναι σχεδόν μείον. Γι' αυτό και ζητώ την κατανόησή σας, γιατί το πρόβλημα αυτό είναι πολύ λεπτό, πολύ ευαίσθητο και φυσικά χρειαζόμαστε και κονδύλια. Και εκλυπαρώ και την υπομονή σας. Είναι το ελάχιστο που σας ζητώ αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτοί που εφαρμόζουν τις αποφάσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, τουλάχιστον εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμμετέχει καν στο Ίδρυμα. Ευχαριστώ και ο κύριος Αλαφράκη και εγώ σας προσκαλούμε ε, να ποζάρουμε όλοι από κοινού στην οικογενειακή ιστορική φωτογραφία. Μετά σα υπενθυμίζω ότι έχουμε συνέντευξη τύπου και το γεύμα είναι ελεύθερο. Ευχαριστώ, λύεται η συνεδρία.